Παρακαλώ, καθίστε. Το κακό είναι ότι ε, δεν κάναμε ακόμα τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Τώρα έχω περισσότερους τους εδώ, ε, γιατί δεν ήθελα να κάνω τις ανακοινώσεις της Προέδρου όταν ήταν άδεια η αίθουσα. Να πω καταρχάς ότι η Ευρωπαϊκή ε, Κοινοβουλευτική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που λαμβάνει η χώρα από τις 28 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες ε, θα επιτρέψει σε διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σε τομείς ε, της ε, αρμοδιότητάς τους, κατά τη διάρκεια των οποίων εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την έρευνα της Κομισιόν για την ετήσια ανάπτυξη και τους προϋπολογισμούς. Η συμμετοχή των Ευρωβουλευτών είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε ε, να διασφαλίσουμε ότι θα είναι επιτυχής οι συναντήσεις και θα προωθηθεί το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν αρκεί να έρθετε για δύο λεπτά να υπογράψετε και να εξαφανιστείτε. Τώρα για τις τριμερείς, για, τους, ε, για τα θέματα του ενιαίου Μηχανισμό Εποπτείας 16 Ιανουαρίου. Παρακαλώ λίγη ησυχία, υπάρχουν πολλοί ψήφιροι μέσα στην αίθουσα. Να σταματήσω λίγο να μιλάω μέχρι να ηρεμήσετε. Ωραία. Η εξέταση του θέματος ε, ε, για την ΕΤΑ και το ECB, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επίσης ε, ε, προχωρούν. Έχουμε στις 23, 24 και 28 Ιανουαρίου συναντήσεις για την οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και για τον κανονισμό. Έχουμε τρεις πολιτικούς ε, τριλόγους. Ε. Στις 10 Ιανουαρίου συζητάμε θέματα όπως τα συγκρίσιμα κριτήρια, μέτρηση κινδύνων, διαχείριση κρίσεων, Επίσης ε, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αποκάλυψη πληροφοριών με βάση τα γραπτά σχόλια των συμμετοχών στις τριμερίς ε, και στις 28 Ιανουαρίου εταιρική διακυβέρνηση και η επόμενη τριμερής είναι στις 30 Ιανουαρίου. Επίσης να θυμίσω σε όλους τους χιώδεις ότι πρέπει να αναφέρουν οποιασδήποτε διμερείς συζητήσεις έχουν με την Ιρλανδική Προεδρία. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα. Υπάρχει μια τάση να γίνονται διμερείς συζητήσεις για τις οποίες εγώ ως πρόεδρος δεν γνωρίζω τίποτα, για τις οποίες άλλα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας δεν γνωρίζουν τίποτα και να μην χάνουμε χρόνο ε, να έχουμε κάθε φορά ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη των τριμερών που να αναφέρεται σε διμερείς συζητήσεις που οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν. Θα σας, σας λέω ότι θα το βάλω στην ημερήσια διάταξη αν τελικά δεν, δεν ξέρουμε τι συζητείτε εκ των προτέρων. Επίσης, ε, να σας πω ότι έγραψα ήδη στον νέο πρόεδρο του Eurogroup και του ζήτησα να έρθει για συζήτηση με την Επιτροπή και να συνεχίσουμε στα ίδια πλαίσια που είχαμε ξεκινήσει με τον Ζαντ Κλοντ Γιούγκερ, με τον οποίο είχαμε πολλές ικανοποιητικέ συζητήσεις. Τέλος, οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας θα λάβει χώρα στις 5 σήμερα, με τον κύριο Μάικλ Νούναν, στην Επιτροπή μας. Σε περίπτωση που τελειώσουμε νωρίτερα τις ψηφοφορίες, να θυμάστε ότι στις 5 πρέπει να επανέλθετε. Σας το ξαναθυμίζω. Φυσικά η εναλλακτική είναι να τραβήξω τις πληροφορίες μέχρι τις 5. Ή εσείς να το κάνετε. Βάλτε τις κάρτες σας στο μηχάνημα για να κάνουμε ένα τεστ πρώτο. Ζαν Πολ, κάτι θες να πεις. Θα έχουμε ένα δίσκο... Δύσκολο θα είναι το απόγευμα με την ψηφοφορία. Ο κύριος ε, Σικλώνα από την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος είναι μαζί μας, τον χαιρετήσω. Να δω, με βάση το, τι, το πόρισμα της ε, ψηφοφορία θα αποφασίσουμε ότι θα τον κρατήσουμε, να το στείλουμε πίσω στους σοσιαλιστές μπαλάκι. Έχουμε την κάτα του, όχι τον ίδιο. Madam Chair, <laughs> Madam Chair. Α <laughs> une décision des huissiers, je crois. Ας τον ρωτήσουμε πώς αισθάνεται. Μα δεν είναι εδώ, κύριέ μου. Α, πολύ ωραία να κοροϊδεύουμε όταν λείπει κάποιο. Κάνουμε τη αστεία και όταν λείπει κάποιο. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε αυτή την δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. Please do test, because occasionally... No. We have one too many green. Έχουμε ένα πράσινο παραπάνω. Ακόμα και τώρα. Right. We've got two more buttons to be pressed. Άλλα δύο κουμπιά, άλλα τρία κουμπιά πρέπει να πατηθούν. 49 ε, βάλαν την κάρτα, 41 άτομα βάλαν την κάρτα τους, αλλά έχουμε 39 ψήφους. Υπάρχει κάποιος που πάτησε το, το κουμπί αλλά δεν άναψε το φως. Είναι προβληματικό όταν βάζουν 41 άτομα την κάρτα τους αλλά δεν βγαίνουν 41 φώτα. Α, τώρα είναι εντάξει όλα. Ψηφίζουμε πρώτα την έκθεση της 22ης ετήσιας έκθεσης τη Ε, συμβασμός 1, υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, υπέρ, κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν άκουσα. Vote's closed. Πέρας 24 υπέρ, 17 κατά. Ε, περνάει. Συμβασμός Β. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός C. Γάμα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά. Ξαναψηφίζουμε τη 42. Υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Ακόμα ένας. Ψήφισαν όλοι. Κάποιος δεν πάτησε το κουμπί του, αλλά εγώ κλείνω τώρα την ψηφοφορία. 23 υπέρ, 18 κατά. Δίκιο είχα. Συμβιβασμός D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός E. Υπέρ. Α, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Το δεύτερο τμήμα του συμβασμού Ι. ε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Come on, more to, more to vote. Three more, three more buttons to press. Two more, one more. Thank you. Ακόμα τρεις. Ωραία, ολοκληρώσαμε την ε, ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά και 20 υπέρ. Συμβασμός F σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αλλά θα το ελέγξω. Νομίζω ότι εγκρίνεται, θα το ελέγξω. Ακόμα πέντε πρέπει να πατήσετε το κουμπί σας. Ακόμα τρεις. Ακόμα δύο. Γιατί κλείνω την ψηφοφορία γρήγορα. Εγκρίνεται 23 υπέρ, 18 κατά. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 3. Σε ένα τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Γκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Υπέρ, υπέρ, ακόμα. Εγώ έχω στη λίστα μου το 76. Θέλουμε να ψηφίσουμε χωριστά το 76. Δεν καλύπτεται από το συμβιβασμό. Έτσι, σωστό δεν είναι αυτό. Ψηφίζουμε λοιπόν την 76. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Συμβιβασμό H. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός I υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκανα λάθος για την ε, τροπολογία 58. Μα να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ah, check, and that is Απορρίπτεται, όπως λέει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, δεν, φταίει το, δεν φταίνουν τα μάτια μου. συμβασμός J. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές ελέγχω την 75 γιατί νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιος κερδίζει. Ψηφίστε ακόμη οι τέσσερις που δεν έχετε ψηφίσει, τώρα πιέζοντας το κουμπί σας. Κλείνω την ψηφοφορία. Τελευταία ευκαιρία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 ψήφου υπέρ, 23 κατά. Συμβασμός L υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός M υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα θα το ελέγξω. Ε, νομίζω ότι μόνο το, το Λαϊκό Κόμμα και το ECR που δεν είναι πλειοψηφία ήταν υπέρ. Ακόμα ένας δεν έχει ψηφίσει. Κλείνω την ψηφοφορία. 24 in favor. 24 υπέρ, 20 κατά. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ο επόμενο συμβασμό σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ. Μπερδεύτηκα. Θα το ελέγξω γιατί μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαφής πλειοψηφία. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ ψήφισε. Παρακαλώ κάποιος να βγάλει την κάρτα του. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 19 υπέρ, 25 κατά. Συμβασμός ο, ου, όμικρον, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μόνο το έλκα ψήφισε διαφορετικά, δεν χρειάζεται να το ε, ελέγξω. 89 υπέρ, κατά, αποχές θα το ελέγξω. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Νομίζω. Αυτός ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 παρομοίως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 114. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός R σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός T υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ και όλες οι άλλες διαγραφές κατά αποχές εγκρίνεται Πού είμαστε τώρα Συμβασμός 2 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός V1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός V2 υπέρ Παρακαλώ για τον V2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός X σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Πρώτο τμήμα του X. Υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τον, το υπόλοιπο έχει νόημα. Το δεύτερο τμήμα δεν έχει νόημα, από ό,τι φαίνεται, αφού απορρίψαμε το πρώτο τμήμα. Αλλά το τρίτο τμήμα έχει νόημα. Συμφωνεί ο εισηγητής, ναι. Υπέρ του τρίτου τμήματος, κατά χές εγκρίνεται το τρίτο τμήμα. Να το εγκρίνω ηλεκτρονικά, εφόσον θέλετε. Ακόμα τρεις να έχουν ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ, 21 ψήφους κατά. Πάμε στις διαγραφές. 152 και λοιπές. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Νομίζω, αλλά θα το ελέγξω. Ένα δεν ψήφισε. Ψηφίστε. Εγκρίθηκε τελικά. 28 υπέρ, 16 κατά. Πάμε στο συμβασμό Y. Υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. Συμβασμός Z. Συμβασμό Z. Και δεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκατόν και τις υπόλοιπες διαγραφές. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο συμβιβασμό ΑΑ σε δύο τμήματα. Ελα... What about 163? No, it says four. Compromise AA, all those in favor. Αλφα, αλφα. Πι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ήταν το πρώτο τμήμα, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το πρώτο τμήμα του ΑΑ. Νομίζω ότι απερίφθη. Αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Vote if closing the vote. Απορρίπτεται, ναι. Με 18-27. Και τώρα θα ψηφίσουμε αυτά είναι τις, διαγραφές 66 και 166 και λοιπά, ποιοι είναι υπέρ, και λοιπά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και τώρα πάμε στη συμβαστική το Β, αλλά έχει από ΑΒ έχει όμως αποσυρθεί και πάμε προ 172 και τις άλλες σχετικές. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 175 και 176. Είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εσύ, συμβαστική εσύ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ. κατά αποχές Εδώ πέρα τούτε η ψηφορία, γι' αυτό εγκρίνεται. 24-19. Ε, AD, συμβαστική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AE, αε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AF, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AG, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 έχει αποσυρθεί. Καλώς. Πριν προχωρήσουμε, στο 203 έχουμε μια προφορική τροπολογία. Εδώ είναι στη θέση μου λένε. Εδώ λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν θα πρέπει να εμπλακούν επίσης ώρες και με της υγιής αρμοδιότητας. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Συμφωνείτε? Ναι, ωραία. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 καταπίπτει και πάμε στο 204. Υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται J σε τρία τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Θέλω να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσανε όλοι. Όμως ψήφισε ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ψήφισαν όλοι πέρασε. Εγκρίνεται 23-21. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Σε δύο τμήματα το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλει το λόγο ο εισηγητή. Η εισηγήτρια. Η Θέλετε να αλλάξουμε για το 2. Ματία. Αφού εγκρίθηκε η συμβαστική, δεν έχει νόημα. Εγκρίθηκε ο συμβασμό εκτό από το κομμάτι που, προέ... που περιέχεται στο δεύτερο τμήμα. Εκεί που λέει, που λέει EMU ε, θα ε, Αυτό ψηφίσαμε. Δεν συμβαστική τροπολογία όμω, λέει η κυρία ματίας Ήταν το πρώτο τμήμα λέει πρόεδρος. Ματίας. Μα το πρώτο τμήμα είναι η συμβαστική. Όχι, όχι δεν ισχύει αυτό λέει πρόεδρος. Όλα αυτά εκτός από το κομμάτι που μας είχε βρει να διαφωνούμε θέλουμε να ανασβήσουμε και που λέει στα πλαίσια αυτού του χάρτη πορείας για ένα αυθεντικό κλπ. κλπ. Αυτό είναι το τμήμα υπερφών Το να μην έχουμε τη φράση που διαβάσατε. Αν ψηφίσετε πέρα δηλαδή θα μείνει αυτή η φράση. Αν ψηφίσετε κατά σημαίνει ότι αυτό το οποίο διαβάστηκε θα διαγραφεί, θα απαλληθεί. Επομένως όλοι όσοι είναι υπέρ της φράσης αυτής, ε, ε, χάρτη πορείας για ένα ε, αυθεντικό υπέρ κατά αποχές, επομένως λέξει. λέξεις. AL, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 204. Τις δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κάτω. AM, το δεύτερο τμήμα, δεν το έχετε. 241. 241 λέει ο κ. Όχι, το 241 και το 246 έχουν καλυφθεί από το AL, αλφα λάμδα, το AL. Λέει πρόεδρος, καλώς. Και ψηφίσαμε υπέρ του πρώτου τμήματος του AM, υποφορές της γυναίκες. Οπότε τώρα, σχόλια. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.36 Υπέρ Κατά Ελεκτρονικός έλεγχος για το 2.36 Άλλοι τρεις, άλλοι δύο. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 18-27. 2-43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2-44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2-45. Υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά πρέπει να κάνουμε έλεγχο Άλλοι πέντε πρέπει να ψηφίσουν. Άλλοι δύο. Ευχαριστώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 21-24. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη τροπολογία. Τρία κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Άλλοι δύο να ψηφίσουν. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τελική παράγραφος γάμα. Συ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. Δέλτα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. το Τροπολογία 8. Υπέρ. Abstentions carried. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Έχω αντιφατικά μήνυμα του ΕΛΚ για το 9. ποιο είναι υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται, νομίζω. Αλλά ας κάνουμε καλύτερα έλεγχο. Votes closed. It is carried, 2718. Sorry, it looked closer than that. Uh, 11, all those in favour. Against, abstentions, rejected. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της ιδιωτικής AIDS Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 16. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Αποχές. Αλήθεια πρέπει να ψηφίσουν. Άλλος ένας, πέρας. Εγκρίνεται. In favor. 18. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Τα αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 22 υπέρ. Αποχές. Απορρίπτωτα. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε ελληνική ψηφορία για να γίνει τελική ψήφιση. Okay, it's every voted, votes closed, and that is carried. 23 in favour. Εγκρίνεται 23-22 χωρίς αποχές. Πολύ σαμπραστική ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. trying to move on to the EIB report, but I haven't got a voting list. Sean, just one thing. There's uh, an addition after the Right, we've got... Um... Α, μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ακόμα μια χωριστή ψηφοφορία που θα σας την εξηγήσω όταν έρθει η ώρα. Όμως τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμβαστική ε εις 2 τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο 16 εις 2 τμήματα, πρώτο τμήμα, Α, για συμπαθάτε με, πρόεδρο, γιατί παρέλειψα τη συμβαστική F. Εγκρίνεται. 16, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πρώτο τμήμα του 16.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 abstain. I can't cope with this chatter and absence of hands, so we'll check. Και ψηφίζετε και δύσκολα τα χέρια σας. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα τώρα. Votes closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 14.30. Συμβαστική G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Βαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ 21 κατά Ας κάνουμε έλεγχο για το 21. Άλλοι τέσσερις. Άλλοι τρεις, άλλοι δύο. Πέρασε ο τώρα είναι αργά, εάν δεν ψηφίσατε. Και απορρίπτεται 18-25. Το αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ, κατά εποχές. Εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα λέει ενισχύει τη σημασία του προοδευτικού βάρος της ΤΕ κλπ. Το δεύτερο είναι η θεωρία ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΕΤΕ να διατηρήσει την αξιολόγηση ε, του τριπλού αλφα. Πρώτο τμήμα, που είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα, που είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Κόντ. Τρία. Υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Κόντ. 7. Πέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. One more to vote. Vote's closed. Άλλος ένας πέρασε. Ingredient. Κοντ 8. Πέρα. Παρακαλώ, περισσότερα χέρια και λιγότερη κουβεντούλα. Είναι πιο γρήγορα. 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κοντ εννέα. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Κοντ δέκα. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Κοντ 11. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Εδώ λέω ότι καλύπτεται όμως από, την, από το U, τη συμβαστική U. ψηφίζουμε, αλλά θα κατησχίσει το ίδιο εάν υπερψηφιστεί αργότερα. Επομένω, αυτή θα, το αποτέλεσμα τη συμφορία έχει προσωρινή ισχύ. 24 επομένω. Υπέρ, κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Αφού απορρίπτεται τόσο το καλύτερο κατά κάποιο τρόπο βολεύει. 25. Και αυτή το αποτέλεσμα θα έχει προσωρινή ισχύ. Υπέρ κατά και εγκρίνεται εγκρίνεται, αλλά ίσως κατησχίσει το χείο. Αν το ίδιο και στο 26. Εξαρτηθεί τι θα γίνει με την ε, πρώτη μήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουμε ψηφίσει αρκετή, οπότε πρέπει να κάνουμε ε, έλεγχο. Άλλος ένας Δεν Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική και υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι, αρχικό κείμενο, εγκρίνεται συνοστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το 34 καλύπτεται. Πάμε στη βαστική M. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πολύ περίεργη αυτή η λίστα Πάμε τώρα στο N. Νι. Στο νι, αλλά δεν το βρίσκω. Α, εκεί πέρα είναι. Μερικέ σελίδε πιο κάτω. Δεν έχουν αριθμό άκουσαν σελίδε. Μπορώ να σα πω σε ποια σελίδα είναι. Νι. Συμβαστική νι. Εν, N νίκος. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Και πάμε τώρα στη συμβαστική όμικρον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Πι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Κιου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 46. εγκρίνεται. Όχι, όχι. Πάει το 46 γιατί ψηφίστηκε το μη. 47 εγκρίνεται. Ε, εάν εγκριθεί το J, το 48 θα καταπέσει. φανταστική χ. Γιατί τώρα έχουμε, εάν η χ περάσει, κάποιες θα καταπέσουν. Η 51, υπέρ. Η 51 και αυτή έχει προσωρινή ισχύ, είναι λίγο ε, παράδοξη. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω, όλοι τα λέτε στα αγγλικά, αλλά ε, εάν ήταν εύκολο να τα λέτε πιο απλά γιατί είναι στα αγγλικά, δεν έχει αύξηση τον αριθμό σελίδε. Αυτά πρώτα δεν μπορούν να τα μεταφράσουν οι μεταφραστέ. Τι να σα πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά. Μα βάζετε δύσκολα, μα κάνετε σαμποτάζ, λέει ο κύριο Γκοζέ. Um, ναι, σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτη για μια τροπολογία την οποία την ψηφίζουμε, αλλά, αλλά θα καταπέσει ενδεχομένως όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας του X, του Χ. Του Έτσι, αυτή είναι η σειρά, είναι λίγο ανορθόδοξη. Θα δείτε τι εννοώ. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε το Χ. Λυπάμαι, είναι όλα ανάποδα, αλλά... Να κάνουμε μια κατεξοδότηση πράξη σε σχέση με το πώς θα ψηφίσουμε και μετά να το αλλάξουμε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το ζήτησα, λέει ο Πρόεδρος αλλά κάθε έκθεση είναι διαφορετική. Πάντως ε, το διασκεδάζουμε τουλάχιστον. 51 υπέρ. Έχετε δει το λόγο. Δεν, δεν ψηφίσαμε, λέει ο μιλητής, λέει ο κύριος Ρικέ, το αρχικό κείμενο που αντιστοιχεί στην παράγραφο 11. Ψηφίσαμε το J, Z και άρα κατα κατά 48 και 49 και έπρεπε να, να ψηφίσουμε την, το αρχικό κείμενο της παραγράφου 11. Ό,τι μου λένε, λέει πρόεδρος, το αρχικό κείμενο και εκείνο καλύπτεται από την συμβαστική. Εντάξει. Δεν το λέει στη λίστα. Αλλά τα περιεχόμενα του 11 καλύπτονται από τον J. Πάμε τώρα στο 51. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ρο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. τέσσερα. Συμβαστική S. Εγκρίνεται. Κόντ. Περθμόν 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κόντ 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίτες Αρχικό κείμενο του 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υ Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κόντ 14 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. Κόντ 15 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του 18 υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά Δεν έχει καθόλου το αποτέλεσμα έλεγχος. Τελευταία ευκαιρία πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21-12. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε προφορική τροπολογία από τους πρασίνους σε σχέση με την συμβαστική δι. Τη δεχόμεθα. Κανείς δεν έχει ένσταση. Do we, should we vote, let's vote the oral amendment separately because I think people are a bit... Να την ψηφίσουμε χωριστά γιατί επικρατεί κάποια σύγχυση. Vote the Greens oral amendment. Πρώτα πρώτα την προφορική των Πασίνων. Τι είναι υπέρ της ε, προφορικής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέρας. Απορρίπτεται η προφορική. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική δι χωρίς την προφορική τροπολογία. Περ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. This. That's all covered. We... What's covered? 70. Okay, we're going to amendment 70. Πάμε στο 70. Αχ, μισό λεπτό. Συμπάθατε με, διότι ψηφίστηκε το Β σαν να μην ήταν κατά διέρεση, με χωριστή ψηφορία. Επομένω, ε, να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί το πρώτο τμήμα και κατόπιν το δεύτερο, εκεί που περιέχονται οι λέξεις, η φράση this word, these words. Θα δούμε κατά πόσον θέλουμε ή όχι να γίνει αυτή η υπενθύμηση, recalls. Υπέρ κατά αποχές γίνεται. Συγγνώμη για τη σύγχυση που σας μπέρδεψα. Done the oral amendment that, that αλλά δεν κατάλαβα ότι η προφορική τροπολογία είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Άρα να κάνουμε τώρα την ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Για το πρώτο εννοεί. Προφανώς πρώτος που λέει μη Μυθιλής 13. Right, one more to vote if you're voting. Okay, vote's closed. Second part. One more person to vote. If you're, are you all happy? Right. With... Άλλος ένας, ευχαριστημένοι, τέλος. Απορρίπτωτα. Πάμε τώρα στο 70. κατά αποχές εγκρίνεται. 72 δύο υπέρ. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική χ. Εξ Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κολτ 16. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Αναπολύπτεται. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. Συμβαστική β. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οκτώ εγκρίνεται και το οκτώ. συμβαστική C εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφορία τώρα για το τελικό κείμενο. I think you have the pages numbered. Yeah, right. The thing is, it's the, the hot water loose parts. And that is carried 37 in favor no against and 5 abstentions. 37-0 με 5 αποχές. Συγχαρητήρια. η συγχαρητήρια που τα βγάλαμε πέρα με αυτή την, την μπερδεμένη μορφή τη έκθεσης. το λόγο. Μετά από αυτή την εμπειρία, έτσι σε ε, πνεύμα καινοτομία. Θέλετε την επόμενη φορά να έχουμε μια λίστα ψηφοφορία και να πηγαίνουμε μια πάνω μια κάτω. Και αυτό μπορεί να γίνει κάποια μέρα. Πότε δεν ξέρεις. Το 16 αναβλήθηκε.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 Έκθεση Κάζα. Να ψηφίσουμε όλες μαζί τις 3, 4, 21, 22, 23 και 25. Αν έχουμε Όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές. Εγκρίνεται. 25, 26 αποσύρονται. Α υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Όλες τις συνδυάμεσεις τώρα. 28 μέχρι 8 όλες μαζί όσοι είναι υπέρ είναι κατά εγκρίνεται β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ αποχές εγκρίνεται σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 με 20 στο τέλος, είναι υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται και θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφορία για το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε. Άλλος ένας να ψηφίσει. Πέρας. 41.00. Ψήφισμα τώρα. Ψηφίζουμε. Κάποιος το βάζει και το βγάζει. Μήπως είναι καλύτερα κάποιος να το κάνει επίτηδες και θα είναι χειρότερο άμα είναι χαλασμένο το μηχάνημα. Άλλοι τρεις. Άλλος ένας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που βοηθήσατε να το κάνουμε μια ομαδική ψηφορία που βοήθησε τόσο. Okay, right. Uh, let's all settle down. Time to panic again. Um, we now have uh, the draft report. Τώρα έχουμε το σχέδιο έκθεσης της Λίζας Φερέρια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με την Ατροπολογία 120. Ξεκινάμε. Εδώ. Περ. Συγγνώμη, αν υπάρχουν συζητήσεις, δεν μπορώ να κάτσετε παρακαλώ και μετά βλέπουμε. I assume everybody what they're doing. We are now going to attempt. Ωραία, αφού καταλάβατε τι κάναμε, θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε πάλι την 120 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Άλλο ένας θα ψηφίσει, κλείνουμε την ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία κάποιο ε, δεν ψήφισε. 22 υπέρ, 18 κατά. Χωριστή ψηφοφορία Συμβασμός α πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Στην 128 πρώτα αυτή θα κάνουμε. Μόνο για το παραγωγικό σύνολο. Ναι προφορική τροπολογία φαίνεται ότι ε, μάλλον βάζουμε τη λέξη μη παραγωγικό σαν productive. Αν είστε υπέρ θα την ψηφίσουμε χωριστά υπέρ. Κατά. Αποχές. Φίλιπ, νομίζω ότι καταψήφισε τη δική σου προφορική τροπολογία, αλλά εγκρίνεται ούτως ή άλλως. Αυτή αντικαθιστά την 128, οπότε πάμε στην 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα τι έκαναν οι άλλοι, οπότε θα το ελέγξουμε λίγο. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, δεν σας βλέπω. Πρέπει να ελέγξουμε. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν. Αν ψηφίζετε. Άλλος ένας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 132. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γι' αυτό πάμε στην 133. Υπέρ. Που είναι διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 143 λοιπόν. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία C σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός D, υπέρ. Κάπως να ψηφίζετε μαζί οι ομάδες. Ξανά συμβαστική D, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική Ή e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός F σε δύο μέρη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία G Yes. Εκτός μικροφώνου. Ξέχασα να πω ότι θέλαμε να ζητήσουμε προφορική τροπολογία εδώ. Στην ουσία είναι απλώς η υποκατάσταση της λέξης severe economic downturn. Σοβαρή οικονομική ύφεση αντί για exceptional circumstances, εξαιρετικές περιστάσεις. Κατά ε, δεν χρησιμοποιήθηκε η λέξη που υπάρχει στο εξάπτυχο, στο six pack. Είναι λοιπόν μια προφορική τροπολογία η Κομισιόν να εξετάσει την κατάσταση των κρατών μελών υπό το φως ε, της σημαντικής οικονομικής ε, ύφεσης αντί για τις εξαιρετικές περιστάσεις. Γιατί η αναθεωρημένη έκθεση δεν χρησιμοποιεί ε, το exceptional circumstances, αλλά το τον άλλο όρο που ανέφερα. Αυτό είναι στα πλαίσια μιας συμβαστικής λύσης που συμφωνήσαμε έτσι ώστε να έχουμε τα όσα γράφει το νομικό κείμενο και όχι αφηρημένες έννοιες όπως το εξαιρετικές περιστάσεις. Is this what I'm sorry, Συγγνώμη, δεν καταλάβαινα τι λέγατε ότι πρέπει να μπει και τι ε, πρέπει να βγει. Είπατε κάτι για το εξάπτυχο, για το δέσμι των μέτρων. Να το επαναλάβω. Συμβαστική τροπολογία F. Είναι απλό έχουμε συμφωνήσει. Καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη υπό το φως των εξαιρετικών περιστάσεων. Όπως ορίζεται στην αναθεωρημένη SCP. Προτείνουμε υπό το φως των εξαιρετικών περιστάσεων αυτή η έκφραση να αντικατασταθεί από το Severe Economic Downturn σοβαρή οικονομική ύφεση. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί το κείμενο. Καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη υπό το φως της οικονομικής, ε, ε, σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως αναφέρεστε στην αναθεωρημένη SGP. Κυρία Πρόεδρε, εγώ το κάνω ναι, ο συμβασμός, αλλά ο Σκιώδης δεν μας είπε ακριβώ τι είναι αυτό που συμφωνήθηκε στο συμβιβασμό ή λίγο πολύ. Δεν ξέρω ακριβώ τι θέλουν να κάνουν οι άλλοι, αλλά ψηφίσαμε. Αν αρχίζουμε να βρίσκουμε άλλες διατυπώσεις, δεν είναι και πολύ θετικό για την ποιότητα της δουλειάς μας. Κοιτάξτε, ψηφίσαμε και απορρίψαμε το να αλλάζουμε τις λέξεις για να ε, συμφωνεί με κάτι άλλο δεν αλλάζει τίποτα σε επίπεδο κειμένου, ας ξαναψηφίσουμε. Αυτή είναι μια αλλαγή στο κομμάτι που πέρασε, μάλλον. Ήταν στο πρώτο κομμάτι, Ζαμπόλ. Απορρίψαμε το δεύτερο τμήμα. Εντάξει, ξεχάστε το. Αν είναι μεγάλο το θέμα, το ξεχνάμε. Για άλλα 10 δευτερόλεπτα, αν περιμένετε, θα το λύσουμε. Στο σημείο, στο πρώτο κομμάτι που υπερψηφίσαμε, Ζαμπολ, υπό το φως των εξαιρετικών περιστάσεων αναφέρεται, αλλά το exceptional circumstances θα πρέπει να γίνει severe economic downturn. Εντάξει. J'ai un problème parce Εγώ έχω πρόβλημα, όπως και ο συμβουλός μου. Γιατί μιλάμε για το 1 ή για το 2. Για το 1. Πριν μας μιλήσατε για το 2. La deuxième est rejetée. C'est celle qui a été votée. bien rejeté. Ma proposition, c'est Et il n'y a pas dans le SPG le. εκτός μικροφώνου. Ce qui est, c'est ces exceptions circonstances are called severe economic downturn. Ça, c'est le, le wording VSGP et c'est ça qu'on adresse quand on parle d'exception. Oui, ça, pas de problème. Du moment qu'on parle de la même chose. Κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Νόμιζα ότι δεν μιλούσαμε για το ίδιο πράγμα. It's, it's our voting performance that takes a severe downturn at the moment. Η ψηφοφορία έχει υποστεί σημαντική ύφεση αυτή τη στιγμή severe downturn. Εντάξει, επιβεβαιώνω ότι με την διατύπωση που προτείνει η Λίσα θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Συμβαστική τροπολογία F αναθεωρημένο πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την ε, τροποποίηση της διατύπωσης. Συμβαστική τροπολογία G. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρα πάμε στην 173 υπέρ. Κατά αποχές εκρίνεται. Πάμε στο συμβαστική τροπολογία H δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Ίσως να μπερδευτήκαμε λίγο. Αν είναι να υπερψηφίζουμε γιατί το χωρίσαμε σε τμήματα. Πέρα στις ε, ψηφοφορίες. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην 183. Favor against. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δύο μέρη υπέρ κατά. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για 191. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα. Okay. So I, just I think got to start voting now. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε. Ωραία. Απορρίφθηκε όπως είπα. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 191 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία J. Δύο μέρη, μάλλον τρία. Υπέρ στο πρώτο κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτό 13 υπέρ 13 υπέρ τη Σάφκο. Περιμένω τα ΕΛΚ. Δεν δείχνεται. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μάλλον το δεύτερο μέρος πρέπει να καταπέσει. Από μόνο του δεν έχει νόημα. Πάμε στην 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία M σε τέσσερα μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέταρτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2-2-1 υπέρ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νέα συμβαστική τροπολογία O. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 233, μάλλον τη 234. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 236 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 238 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 242 υπέρ 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 με προφορική τροπολογία από τους πράσινους. Πρώτα, λοιπόν, ψηφίζουμε και για την προφορική τροπολογία. Ελέγχει Ζαμπόλ. Λαμβάνει υπόψη την ε, θέση σε ισχύ. Okay. Two, 243 with the amendment. 243 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 244 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Q υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία R σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. I think I'm supposed to be voting now. Has everybody voted? Votes closed. Ψήφισαν όλοι υπέρ τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 22 με 19. 258 υπέρ. Υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 262 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 263 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία από εμένα και τον εισηγητή τη συμφωνήσαμε με την Επιτροπή Απασχόλησης για να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αύκο 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μια νέα... Ένα νέο υποκεφάλαιο από κάποιον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κι άλλη μία ε, υποκεφαλίδα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. These go in, so we now go down to budget Budget... Πάμε στο προϋπολογισμό 6 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμός 11 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 4 περιμένετε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και άλλη μία υποκεφαλίδα, περιφερειακές πολιτικές υπέρ, κατά, αποχές. Είναι κανείς κατά της νέας υποκεφαλίδας, εγκρίνεται. Είναι στην κατάλογο ψηφοφορίων να ψηφίσουμε αν μπλοκ μέχρι το τέλος να ψηφίσουμε τις Ρέτζι από το 1 έως το 7. Unblock. Όχι. Συγγνώμη, δεν γίνεται. Ρέτζι 1. Υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 5. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνταγματικές υποθέσεις υπέρ κατά αποχές είναι υποκεφαλίδα. Να κάνουμε την αφικό unblock, όχι δεν μπορούμε. Αύκο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές ε, κατά. Can we take AFCO? Can we take AFCO 3 onwards on block? Από το 3 και μετά μπορούμε να πάμε en block. Ωραία, όλα τα υπόλοιπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Θα κλείσω την ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας. Είμαστε υπέρ της ΑΦΚΟ 24 και κάτω. Πάμε τώρα στην συμβαστική τροπολογία S σε έξι τμήματα. Αν τα βρω. Ένα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερον. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται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 Δεύτερο μέρος. Αυτό απορρίπτεται. Αυτό το είδα και όταν σηκώσατε τα χέρια. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέταρτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέμπτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έκτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. all those compromises have been rejected. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λάθος στην ερμηνεία της, του καταλόγου ψηφοφοριών. Να μας πείτε λίγο ποιο είναι το πρώτο τμήμα, ποιο είναι το δεύτερο στον συμβαστική τροπολογία S. Όχι, όχι, ναι, ναι. These No, look, okay. I've had a request and I will tell you what is in my voting list. It says... Έχω ε, το εξή αίτημα. Το, σημείο, το τμήμα 1 είναι μία σύσταση χωρίς τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω. Και τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω είναι πρώτον, το πρώτο κομμάτι της σύστασης 1, το δεύτερο τμήμα της σύστασης 1, οι λέξεις, namely due, οι λέξεις, ε, η φράση που ξεκινάμε with the ECB και η φράση που ξεκινάει in the EU and in the Eurozone in particular. So that's, that's, we voted as we... Όπως θέλαμε ψηφίσαμε, φαντάζομαι, έτσι. Περνάμε τώρα στη συμβαστική τροπολογία τι κάπου είναι στην σελίδα 19 σε τρία μέρα, μέρη. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της τι. Υπέρ. Κατά. Μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ε, την ε, συμβαστική τροπολογία τη στη σελίδα 14. Well, you weren't voting, but the first part was carried whilst the... Δεν ψηφίσατε, αλλά το πρώτο ε, κομμάτι εγκρίθηκε, ενώ εσείς οι σοσιαλιστές συζητούσατε μεταξύ σας. Δεύτερο τμήμα. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν, αν ψηφίσατε. Πέρας της ψηφοφορίας. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται 32 προς 8. Τρίτο μέρος υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε το τρίτο μέρος, γιατί και πάλι είναι διαφορετικό. Ψήφισαν όλοι. Άλλοι πέντε αν θέλουν. Άλλοι δύο αν μπουν στον κόπο. Υπέρ. Εγκρίνεται. 22 προς 18. Συμβαστική τροπολογία U. Σε 9 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεν μπορώ να το κάνω αν κάθεστε πάνω στα χέρια σας. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υπέρ, στο τρίτο. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σημείο 4, τμήμα 4, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 6. Ελέγχουμε το 5. If you have two more to vote if you're voting. I'm going to close the vote. And that's carried 21 to 19. Part 6 in favour. Against. Abstentions. That's carried. Part 7 in favour. Again. Εγκρίνεται υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Εξαρτάται από το προς τα πού θα πάνε οι άλλοι. Δεν βλέπω αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Ε, τμήμα 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία UA με προφορική τροπολογία από τους πράσινους. Εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε με την προφορική τροπολογία. Ναι, ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία W υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά Αποχές πρέπει να ελέγξουμε τη 14. Has everybody voted? I'm closing the vote. And that's rejected 20 to 20. 20 ε, υπέρ, 21 κατά, ε, απορρίπτεται. Η 15 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Μάλλον. Μάλλον θα το ελέγξω. Δεν είδα. Πολύ καλά τα χέρια. 15. Κάποιες εποχές ε, μας μπέρδεψαν. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές. Μπορώ να ελέγξω τη 19. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 21 προς 19. 20 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 28. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Y. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Three more to vote, two more to vote. Άλλοι τρεις πρέπει να ψηφίσουν. Αν ψηφίζετε, πατήστε τώρα τα κουμπιά σας. Κλείνω την ψηφοφορία. Καταπίπτει 20 προς 20. Πάμε στην τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξω γιατί κάποιοι τώρα δεν ψηφίζουν. 29 ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές θα το ελέγξω. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας δεν βλέπω. Πέρα από το γεγονός ότι δεν είμαστε όλοι εδώ. Άλλοι δύο να ψηφίσουν πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια δεν μπορώ να σας μετρήσω. Συμβαστική τροπολογία Z. Αν θέλει κανείς να έρθει εδώ στη θέση μου, είστε ελεύθεροι. Z, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 36, υπέρ. Ζαμπόλ. Ήθελα να ρωτήσω αν ε, ήταν μια γενική προσφορά η προσφορά σας ή μόνο για τις ψηφοφορίες. Γιατί αυτό θα μας κάνει να σκεφτούμε. Ζαμπόλ, μπορείς να έρθεις και να κάνεις την ψηφοφορία όποτε θέλεις. Ξέρω πως αρέσει πάρα πολύ και πόσο εύκολη σου φαίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 42. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΑ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 43, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην AB, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AC υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 60 υπέρ η AC απορρίφθηκε. Συγγνώμη. Έχω παρασυρθεί λίγο. Τροπολογία 53 υπέρ κατά Αποχές. Είναι πολύ κοντά. Πρέπει να το ελέγξουμε για την 53. Lots more people to vote if you're... Είναι πολλοί ακόμα που πρέπει να ψηφίσουν. Άλλος ένας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 προς 18. Τώρα μπορούμε να πάμε στο 60. Τροπολογία 60 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν το είδα. Θα ελέγξουμε την 60. Πέραση closed. Πέρασε ψηφοφορία. Αγκρίνεται 21 προς 18. Ε, Τροπολογία AD, συμβαστική AD, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 61, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ακούω θόρυβο στα ακουστικά μου. Συμβαστική τροπολογία ΑΕ, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η F υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία x Λέει έτσι, εγώ δεν το πιστεύω. AG μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. AH. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα σε μια προφορική τροπολογία από τους πράσινους ε, για την τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 87 87. Κυρία Πρόεδρε, δεν είπα τίποτα πριν, όμως για άλλη μια φορά έχω μια προφορική τροπολογία που ανακοινώνεται και δεν φαίνεται στην κατάλογο ψηφοφοριών. Το άφησα πριν να περάσει, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε και συνήθεια. Very sorry, I, I was not told you hadn't got it. Συγγνώμη, δεν μου είπαν ότι δεν την έχετε. Εννοείται την προφορική τροπολογία για τους πράσινους στην τροπολογία 86. αλλάζει τη λέξη is reflected in στο has an impact on. Δείχνει ένα κενό ανταγωνισμού μέσα στην περιοχή του ευρώ που έχει επίπτωση στις ε, διαφορές ε, για τα επιτόκια. Και τώρα έχουμε άλλη μία που είναι προφορική τροπολογία στην τροπολογία 87. Ε, βάζει τη λέξη όταν υπάρχουν ε, μεγάλα επιτόκια σε κάποιες ε, χώρες μέλη, θεωρούνται εν μέρη ε, ότι οφείλονται σε έλλειψη αξιοπιστίας για την διεξαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μου φαίνεται λογικό. 87 με την προφορική. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 88. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AI σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην AJ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 98. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. AK ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία EL υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά, Άλλο να το ελέγξουμε. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ψηφίζονται εδώ ή ψηφίζουν οι ομάδες. two more to vote. Άλλοι δύο πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 22 προς 18. Συμβαστική τροπολογία ΙΕΜ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, Έμιλη. Σύντομα. Νομίζω ότι η ψηφοφορία αυτή έδειξε πολύ καλά ότι ε, ήταν λίγο περίεργη διαδικασία και γι' αυτό καταψηφίσαμε και η Επιτροπή πρέπει να ε, εξετάσει τις επιπτώσεις για το μελλοντικό ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη για να καταλήγουμε με ένα τέτοιο κείμενο που πηγαίνει προς διάφορες κατευθύνσεις και νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο χρόνο για ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις και να μην έχουμε καθένα την άποψή του έτσι και να την διατυπώνουμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό να είναι σωστή διαδικασία, πρέπει να το δηλώσουμε απερίφραστα και πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνήθως πριν την ψηφοφορία δεν ξεκινάμε ε, να κατακρίνουμε αυτούς που δεν ψήφισαν όπως θέλουμε εμείς. Ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει στη δημοκρατία. Θεωρώ παράδεκτο πριν από την ψηφοφορία να έρχεστε και να λέτε ότι επειδή δεν είχαμε την ικανοποίηση που θα θέλαμε, ε, δεν δουλεύουμε σωστά. Αυτή η ψηφοφορία θα αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία αυτής της Επιτροπής και δεν κάνω κανένα σχόλιο για τη μέθοδο με την οποία έγιναν οι διαδικασίες. Παρατηρώ ότι και πέρυσι είχαμε σε μια, στην προηγούμενη έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είχαμε μεγάλη πλειοψηφία. Και αυτό ήθελα να το δηλώσω. Ευχαριστώ πολύ. Να τονίσω ότι ε, οι επεξηγήσεις ψηφοφορίας έρχονται μετά την ψηφοφορία και όχι πριν. Εγώ επέμεινα να ψηφίσουμε σήμερα γιατί δεν θα πάω στην Ολομέλεια χωρίς θέση της ΕΚΟΝ ξεκαθαρισμένη και δεν θα το αφήσω πλήρω στα χέρια τη Επιτροπή Απασχόληση. Πρέπει να συμφωνήσουμε επί του κειμένου και να έχουμε μια συντονισμένη απάντηση του Κοινοβουλίου εγκαίρω για την Ολομέλεια. Έχουμε λοιπόν κάποιε μέρε ε, για να μπορέσουμε να τα βρούμε μεταξύ των ε, Επιτροπών και μεταξύ μα αν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήδη ήταν θέμα συζήτηση μεταξύ των Επιτροπών, ε, μεταξύ δηλαδή των δύο συγητών. Ευχαριστώ τους πράσινους που σταμάτησαν να παίζουν τον πρόεδρο. Τώρα θα γίνει καταγεγραμμένη ψηφοφορία του κειμένου ως τροποποιήθηκε. Άρχισε η ψηφοφορία. Ωραία. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η έκθεση 19 υπέρ, 21 κατά και καμία αποχή. Okay. Right. Uh, so now uh, in line with the normal... Τώρα, με βάση τη συνήθεια διαδικασία, να σας την πω καταρχήν ποια είναι. Η έκθεση πηγαίνει πίσω στον εισηγητή και το σημείο θα συμπεριληφθεί στο τέλος της ε, συνεδρίασης των τελευταίων συντον... της επόμενης συνεδρίασης των συντονιστών που θα αποφασίσουν τι θα κάνουμε συνεχεία. I will point out that the vote was... Uh, ε, το αποτέλεσμα της φοφορίας ε, επηρεάστηκε πάρα πολύ από την απουσία διαφόρων εισηγητών, έτσι. Πέρασε, πέρασαν ή χάθηκαν τροπολογίες λόγω απουσίας ατόμων. Η συγγήτρια. Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν με συμβιβασμούς και όσοι επέδειξαν καλό πνεύμα συνεργασίας. Δεν θα σχολιάσω όλα τα υπόλοιπα θέματα. Η στιγμή που ζούμε αυτή τη, ε, στην Ευρώπη είναι αρκετά σοβαρή. Νομίζω ότι οι πολίτες μας περιμένουν ένα σαφέστατο μήνυμα προς την Κομισιόν. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να διαπραγματευτώ και να φτάσω συμβασμούς με καλή την πίστη. Αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιδιωκόμενο. Ήτανε, δημιούργησα μηχανίες τη ψυχοφορία. Είχαμε πολλά προβλήματα την τελευταία στιγμή. Ε, τελευταία στιγμή δεν πέρασαν συμβιβασμοί που είχαμε συμφωνήσει. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη δουλειά μου σε αυτό το αποτέλεσμα. Να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί τελικά το Κοινοβούλιο να μην πάρει θέσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών. Ευχαριστώ.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 jean Πολ. Εγώ σας είχα προειδοποιήσει την τελευταία φορά, όταν έγινε το πρώτο σχόλιο για αυτή την έκθεση. Είχα πει ότι οι γενικοί προσανατολισμοί δεν ήταν αποδεκτοί όσοι ε, είχαν από το ΕΛΚ. Ε, αυτά που δεχόταν το ΕΛΚ υπήρχαν στην περσινή ε, έκθεση ήταν αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών από όλε τι ε, πολιτικέ ομάδε. Και είχα πει ότι αν θέλαμε κάτι πιο σοβαρό, χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο. Ε, πέρυσι χρειαστήκαμε πολλέ συνεδριάσει για συμβάσμα. Τώρα είχαμε τι χριστουγεννιάτικε διακοπέ, ε, μειώσαμε την προθεσμία και μα είπαν ότι χρειαζόμαστε το οπωσδήποτε την έκθεση για την ολομέλεια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, δεν υπάρχει έκθεση. Η, η Ελίζα ξενύχτησε για, τις, ε, για τους συμβιβασμούς. Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα. Θα μπορούμε να πούμε βέβαια ότι η Κομισιόν δεν μας είχε δώσει όλα τα στοιχεία πιο νωρί. Πέρυσι μας τα είχε δώσει πιο νωρί. Ε, φέτος αδιαφορεί η Κομισιόν για το Κοινοβούλιο. Και είχα πει Καλύτερα να δοθούν 8 μέρες παραπάνω και να έχουμε ένα καλό έγγραφο, ούτω ώστε να έχει θέση το Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν δεν επικυρωνόταν από την Ολομέλεια, θα, υπήρχε αυτή η θέση του α, Κοινοβουλίου. Σήμερα ε, το απόγευμα το ΕΚΟΦΗΝ δούλεψε για, πάνω σε αυτό το θέμα. Για τη δική μας έκθεση λοιπόν αδιαφορεί τα μάλα Είχαμε πει ότι θα πήγαινε η έκθεση στην Ολομέλεια αν καθυστερούσαμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη χρόνου και η καθυστέρηση της Κομισιόν. Επίσης δεν έχουμε και, και πολλές ολομέλειες. Έχουμε ένα οικονομικό διάλογο με τον ε, Ιρλανδό Πρωθυπου... Συγγνώμη, Υπουργό τώρα και ελπίζω οι βουλευτές να παραμείνουν για αυτό το διάλογο με τον Ιρλανδό Υπουργό. Ευχαριστώ.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

Right. Uh, thank you very much. Um, I'm very to, welcome uh, Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση Καλωσορίζω τον Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, τον Μάικλ Νούναν. Θα έχουμε ένα νέο σύστημα τώρα. Θα μας εκφωνήσει μια ομιλία ο Υπουργός για ένα κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πόσο. Πόσο? Δέκα λεφτά. Και συνεχεία θα έχουμε πέντε λεφτά για ερωτήσεις και αποκρίσεις. Αλλά φυσικά, αν ο υπουργό χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω, θα του τον δώσουμε. Ούτως ώστε να γίνει μια καλή ανταλλαγή απόψεων. Μάικλ, έχεις το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει η κυρία Μπόλς. Ε, ήταν μια, πάντοτε μια πολύ καλή φίλη της Ιρλανδίας ε, και πάντοτε είναι πρόσδεκτη. Μας υποστηρίζει σε πολλά ζητήματα που μας αφορούν. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ υπό την αρμοδιότητά μου ως Προεδρεύοντα του Συμβουλίου των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για να σας δείξω το πρόγραμμα της Ιρλανδικής Προεδρίας ε, του ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα να τις τιμή και στην Κυπριακή ε, και την Δανική Προεδρία. Θεωρώ ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα οικονομικά και φορολογικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2013 βρισκόμαστε σε μια καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόμασταν πέρυσι. Έχει βελτιωθεί η οικονομική δραστηριότητα, ο πληθωρισμός ε, φαίνεται βίωνος, υπάρχει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε κάποια κράτη-μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες που κάνανε κράτη-μέλη, βρισκό, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόοδος ε, και στο χρέος ε, κρατών μελών. Αυτό ισχύει και στις χώρες που υπάρχει το μνημόνιο και όπου έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να μπει τάξη στη δημοσιονομικά τους και να είναι πιο βιώσιμα στο σημερινό ΕΚΟΦΗΝ λαμβάνουμε υπόψη την πρόοδο που υπάρχει στην Ιρλανδία. Όμως αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που παραμένουν και ε, η, ανάπτυξη, η εξέλιξη της αγορές συνεχίζει να μας ανησυχεί. Καλό θα ήταν λοιπόν κατά την Προεδρία μας να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα ζητήματα όπως και στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε τη σταθερότητα για να προωθήσουμε την ανάπτυξη, να μειώσουμε την ανεργία, να αντιμετωπίσουμε την κρίση χρέου και να μειώσουμε και το κοινωνικό αντίκτυπο τη οικονομική κρίση. Όπω γνωρίζετε, πέρυσι οι ευρωβουλευτέ ήρθαν στο Δουβλίνο και αυτό είναι άλλη μια δυνατότητα για να συνεχιστεί ο διάλογο μα. Θα έλεγα ότι προσπαθώντα να πετύχουμε την ημερήσια διάταξή μα, το Κοινοβούλιο θα μα βοηθήσει σημαντικά. Η Ιρλανδική Προεδρία αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου ω συνομοθέτη. Είναι καλό λοιπόν να συνεργαστούμε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται. Έχουμε ήδη κάνει καλή αρχή. Κατανοώ ότι υπήρξαν σημαντικές ως τώρα δεσμεύσεις σε πολλά θέματα μεταξύ της Προεδρίας και του Κοινοβουλίου. Ε, θεωρώ ότι ήταν χρήσιμες οι δεσμεύσεις και θα αποτελέσουν τη μήτρα για, τα επόμενα, για το επόμενο εξάμεινο. Ως ε, κοινοβουλευτικοί όλοι έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι θα δώσουμε λύσεις στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Και αυτό θα βελτιώσει την ευζοή όλων των πολιτών μας. Με την βοήθεια αυτού του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε όλες τις προηγούμενες προεδρίες έγινε καλή δουλειά. Εμείς έχουμε την εξή ημερήσια διάταξη. Οικονομική διακυβέρνηση, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Κρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Φορολογία, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η αιτήσια έκθεση ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη το τρίτο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Το βασικό μήνυμα είναι ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές αρχίζουν να δείχνουν αποτελέσματα, μειώνονται τα ελλείμματα, χαλαρώνουν οι εντάσεις, ε, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα σε κάποια κράτη-μέλη συνεχίζει η δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξη έτσι λοιπόν έχουμε πέντε βασικές προτεραιότητες όπως ορίστηκαν στην έρευνα του 2012, όμως διαφορετική είναι η έμφαση, ανεργία και κοινωνικές επιπτώσεις. Αυξάνονται όλα αυτά. Δίνουμε περισσότερη έμφαση λοιπόν στην έρευνα του 2013. Στην πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου, πιο νωρί σήμερα, έγινε μια χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών. Σήμερα στη συζήτηση η Προεδρία έδειξε τις προθέσεις της να γίνουν συζητήσεις στην για τη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας ε, σχετικά με το κοφήν ε, του Απριλίου του 2013. Σήμερα θα ψηφίσουν στο Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο και τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης. Καλωσορίζουμε τα βήματα που έχει λάβει το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη ε, παρακολούθησης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού ε, Ξαμήν. όσον αφορά τη δεύτερη δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης, ε, θεωρούμε ότι σχεδόν έχουμε φτάσει στο τέλος. Υπάρχει ανάγκη για πρώιμη συμφωνία σε αυτά τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ε, τις προσπάθειες για μια γρήγορη συμφωνία επί του κειμένου. Έχουμε δει το προσχέδιο ε, για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση το περασμένο Δεκέμβρη. Ω Προεδρία θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε από αυτού και ε, να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Φαν Ρόμποϊ. Η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων της Τραπεζικής Ένωσης θα, θα διευκολύνουν το να σπάσουν τα δεσμά μεταξύ ε, των, της Ένωσης και των ε, κρατικών χρεών. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνονται προτάσεις με βάση την προθεσμία του ε, Δεκεμβρίου του 2012 η συμφωνία για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που ε, έγινε στις 13 Δεκεμβρίου στο ΕΚΟΦΗΝ είναι ένα σημαντικό σημείο που θα διασφαλίσει την εποπτεία σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο και για την ε, κανονισμό ε, για την ΕΚΤΕ που τροποποιεί τον κανονισμό του 2010 την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και στο ΕΚΟΦΗΝ. Όσον αφορά το πλαίσιο για την εξηγήνωση των τραπεζών, έχουμε μία συμφωνία που πρέπει να την έχουμε μέχρι το 2013 στο Συμβούλιο. Για να γίνει αυτό δίνεται μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα σχέδια εγγύησης καταθέσεων, η Ιρλανδία σχεδιάζει να ξανανοίξει τη συζήτηση για τα θέματα του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού, της οδηγίας για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και της οδηγίας για την ανάκαμψη και εξηγένση των ε, τραπεζών. Θέλουμε να υπάρχει καθαρότητα ε, για αυτά τα θέματα, ειδικότερα για την εγγύηση των, επενδυ... των καταθέσεων. Ελπίζουμε οι συνομοθέτες λοιπόν να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για την ε, οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις 4 πολύ γρήγορα υπάρχει αυτός ο σημαντικός ε, φάκελος, αλλά και ένας επόμενος ε, που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιανουαρίου. Εμείς θέλουμε να προωθηθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να γίνουν πιο αποδοτικές, ε, πιο διαφανείς και να προστατεύουν τους επενδυτές. Εμείς θέλουμε να υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο και να, να υπάρξει σύντομα μια ε, συμφωνία για τη ΜΑΤ και την ΜΑΡ. Ε, υπάρχει μια σειρά τριμερών με το Κοινοβούλιο, ε, όπως επίσης και στο θέμα των καταναλωτών σχετικά με την οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστοσης για τα κίνητα κατοικία. Υπάρχουν προτεραιότητες λοιπόν στις, στους τομείς όπου μπορεί να υπάρχει πραγματική πρόοδος θέλουμε μέσα στο εξάμεινο της Προεδρίας μας να κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές ώστε να φτάσουμε σε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στο θέμα της φορολογίας. Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών συζητήθηκε στο ΕΚΟΦΗΝ και αποφασίσαμε να πάμε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας. Σήμερα το πρωί η Ιρλανδική Προεδρία επίσης προ... ξεκίνησε τις συζητήσεις για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών που είναι γνωστή ως ε, CCCTB και υπάρχουν ε, προτάσεις που θα διευκολύνουν μια γρήγορη και αποτελεσματική απάντηση σε αυτή τη μορφή απάντησης και θα υπάρχει και ένας ε, μηχανισμός ταχείας ε, δράσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλή αντιμετώπιση των αποδεικτικών συναλλαγών και του προγράμματος για την, για την φορολογία. Η Προεδρία επίσης θέλει να ε, προωθήσει την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, ε, να πατάξει την φορολογική απάπτη και την φοροδιαφυγή. Θα προσπαθήσουμε επίσης να βρούμε μια συμφωνία σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην οδηγία για τη φορολόγηση των από αποταμιεύσει. Τώρα για τον ετήσιο προπολογισμό του 2013 ε, θα προχωρήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση, θα προωθήσουμε την ε, απαλλαγή για το 2011 και θα προετοιμάσουμε κατευθυντήριες γραμμές για το 2014 με τις ακατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές. Το πολιετές ε, χρηματοπιστωτικό πλαίσιο επίση είναι σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή ε, είναι η η ε, Προεδρία μας και η 40η ε, επέτειος της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε μία πρακτική και ουδέτερη προεδρία, όπως έχουμε δείξει και στο παρελθόν, και να προωθήσουμε την ημεράσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και όχι των κρατών μελών μεμονωμένα. Θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε με βάση όλα αυτά, λοιπόν, γιατί έχουμε και ένα μητρό επι... επιδόσεων πολύ καλό και θα συνεργαστούμε ε, και με την Ελιθανική Προεδρία στα μέσα του 2013. Ελπίζουμε ότι με τη δική σας ε, υποστήριξη θα επιτύχουμε ε, αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και θα μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ ότι ήδη έχουν ξεκινήσει ορισμένοι πολύ σημαντικοί τριμερείς διάλογοι και έχει σημειωθεί μια κάποια πρόεδρο, πρόοδος. Τώρα το ΕΛΚΑ έχει να κάνει την πρώτη ερώτηση από το ΕΛΚ, λοιπόν, ο κύριος Ζανπόλ Γκοζές. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος των μελών του ΕΛΚ και ο ίδιος προσωπικά θα ήθελα να σας καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή μας, που είναι μια Επιτροπή που δουλεύει πολύ γιατί τα θέματα της δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρα. Ας το θέσω έτσι. Σας καλωσορίζω λοιπόν και ελπίζω μαζί να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη χώρα σας. Είδαμε τι προσπάθειες καταβάλατε, τι αποτελέσματα πετύχατε και νομίζω ότι αυτό είναι και θετικό για την Προεδρία. Είπατε ότι η Προεδρία σας θα είναι δίκαιη, αποτελεσματική, ρεαλιστική και θα ήθελα ακριβώς να κάνω δύο σχετικές παρατηρήσεις. Μια γενική καταρχήν παρατήρηση. Οχτώ χρόνια ανήκω εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και διαπιστώνω ότι οι διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων γίνονται όλο και πιο δύσκολε. Οι θέσει των κρατών μελών είναι άκαμπτε, παγιωμένε και η συζήτηση με το Κοινοβούλιο είναι δύσκολη. Σε μια διαπραγμάτευση όμω ο καθένα πρέπει να κάνει ανοίγματα και βήματα. Ίσως θα μπορούσατε να διευκολύνετε εσεί την κατάσταση. Επίση έχουμε θέματα τα οποία έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό είναι ανησυχητικό. Καταρχά το 2-pack. Εγώ είμαι εισηγητή για το ένα από τα δύο κείμενα. Το κείμενο εδώ και πολύ καιρό είναι έτοιμο, όμω ε, υπάρχουν ε, σημεία όπου περιμένουμε ας πούμε μία δήλωση η οποία δεν ήταν ε, ικανοποιητική. το κείμενο έχει οριμάσει, μπορεί να ψηφίσει, αλλά δεν έχουμε ακόμα μπορούμε να ψηφίσουμε, αλλά δεν έχουμε, κάνει, δεν έχουμε ακόμα την πλειοψηφία. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Θα μας βοηθήσετε την απεμπλακή κατάσταση και Κάτι άλλο σημαντικό για τα κράτη-μέλη και για τους επαγγελματίες ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ε, για την οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά διάφορα πράγματα αμφισβητούνται εκ νέου. Θα ανησυχούσαμε πολύ αν τα αποτελέσματα που πετύχαμε με την ε, Προεδρία Χ αμφισβητούνται από την Προεδρία χ Χ1, από την επόμενη Προεδρία. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεσή σα. Και είπατε εσεί εξάλλου προηγουμένω ότι θέλετε το θέμα αυτό, ο φάκελο αυτό, να προχωρήσει πολύ. Θα ήθελα όμω να μου δώσετε διευκρινήσει για αυτά τα δύο σημεία και για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί η Ιρλανδική Προεδρία. Οι άλλοι συνάδελφοι μου θα σας θέσουν και πιο λεπτομέρειε ερωτήσεις για τις προτεραιότητέ σα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Γκοζέ. Σας ευχαριστώ για τα θετικά σχόλια που κάνετε για την Ιρλανδία. Η προσέγγιση της Προεδρίας θα είναι να προωθήσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα. Και θα παραμερίσουμε τα εθνικά συμφέροντα και τις εθνικές θέσεις όσο έχουμε την Προεδρία. Η επιτυχία μιας Προεδρίας δεν μετριέται με τον αριθμό των τριμερών διαλόγων ή των ολομελιών κτλ. Αλλά πόσα θέματα βοηθάει για να ολοκληρωθούν. Επομένως, το πρόγραμμα εργασίας μας θα το φτιάξουμε με βάση του τι είναι εφικτό, νωρίς μάλιστα, και θέλουμε να δώσουμε και αρκετό χρόνο ε, για τους φακέλους που είναι πιο δύσκολοι. Ας πούμε, το, πολυ... το FTT το βάλαμε στο πρώτο ECOFIN, σήμερα το πρωί, χωρίς ψηφοφορία. Υπήρχε ήδη ειδική πλειοψηφία, αλλά δεν το θεστάραμε. Κανένα δεν είπε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα καταψηφίσει. Επομένως, περνάμε στην επόμενη φάση. Ε, η επόμενη προτεραιότητα είναι το 2-pack. Είμαι απογοητευμένο που βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια μπορώ να σας πω ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε τίμοι ενδιάμεση μεσολαβητές και διαπραγματευτές μιας συμφωνίας. Έχω εδώ τον πρέσβη και θα βοηθήσουμε όλοι ούτως ώστε να πετύχουμε συμφωνία. Διαβάστε το φάκελο. Ε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει κοντά στη συμφωνία. Ο πρόεδρος μας και ο πρόεδρος Μπαρόζο ε, το βράδυ ζήτησαν ευελιξία γενικά, ούτως ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Διαβιβάζω αυτή την δήλωση. Εγώ δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε αυτό το ρόλο. Για την τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος, ε, δίνουμε προτεραιότητα. Ξέρω ότι και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θέλουν να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις επόμενες εβδομάδες. Είναι ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα γιατί πολλά σημαντικά πολιτικά θέματα που δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Επίσης το κείμενο είναι πολύ τεχνικό και περιπλέκει τα πράγματα. Μέχρι στιγμής στην Προεδρία μας έχουμε προβλέψει τρεις συνεδριές ομάδα εργασίας και δύο πολιτικούς διαλόγους. Η ομάδα εργασίας μου λένε ότι έχει προχωρήσει και διάφορα θέματα ε, έχουν κλείσει. Βέβαια υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ε, κατάλογος ανοιχτών θεμάτων ακόμα και πολιτικών. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμφωνία, θα το κάνουμε με... όσε όσες περισσότερες συνεδριάσεις μπορούμε, όσες χρειάζεται, εν και θα στείλουμε υπαλλήλους και αξιωματούχους ε, πολύ ικανούς, πολύ αρμόδιους, με γνώση των θεμάτων στους διαλόγους. Και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και το Συμβούλιο με το μέρος μας. Η Αρλίν Μακάρθη από τους Σοσιαλιστές. Um, και εγώ να σας συγχαρώ ότι είναι παγκόσμιος πρωτοαθλητής η Ιρλανδία όσον αφορά την διαχείριση των οικονομικών της. Δεν ξέρω τώρα βέβαια και στο κοφίν θα έχει θέση και κάποια γυναίκα. Ναι, ναι, μία. Μόνο μία. Όχι. Εννέα, ναι, τότε να τις αθροίσουμε. Ξέρω κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν πάρα πολύ ψηλέ προσδοκίε όσον αφορά την Προεδρία σα και εγώ είμαι 18 χρόνια εδώ και ξέρω ότι κάθε φορά που είχατε την Προεδρία σα ήταν αποτελεσματική, δίνατε σημασία στα αποτελέσματα. Και καταλαβαίνω ότι έχετε ε, τρομερή τρομερή μέσα διάταξη. Να σας πω λοιπόν το θέμα αυτό το οποίο αναφέρατε ε, δηλαδή την κατάχρηση των κανόνων της αγοράς κλπ. Ναι, έχουμε ε, την κρίση, έχουμε τι θα κάνουμε ε, με τη ΣΥΠΑ, για να δούμε θα γίνει με τις κυρώσεις που δεν έχουμε εμεί και έχουν οι Αμερικανοί. Όσον αφορά ακριβώ τη χειραγώγηση της αγορά. Οπότε Λέγαμε ότι αυτό κάτι θα γίνει, το είχαμε πει τον Οκτώβριο, νομίζω ότι θα το κάνει η Κυπριακή Προεδρία, δεν το έκανε, επομένω τώρα έχουμε ποντάρει πάνω σα. Ό,τι μου λένε πάντως, πηγές μου, η Ιρλανδική Προεδρία δεν θα δώσει προτεραιότητα με ε, τριλόγους όσον αφορά ακριβώς την κατάχρηση της αγοράς. Δεν θα δώσει προτεραιότητα στο θέμα, επομένως για πέστε μου, πότε θα έρθει η ώρα ότι αν δώσετε αυτό το πολιτικό ε, μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε στο μέλλον στην Ευρώπη χειραγώγηση της αγοράς. Έχουμε αυτά τα 30 δις για τη διάσωση των Ιρλανδικών τραπεζών. Ε, τότε δεν θα πρέπει κι εσείς κάτι να πείτε στους ε, ε, ψηφοφόρους σας. Να τους πείτε ότι δεν πρόκειται στις συμμετοχομικές υπηρεσίες να ανεχθούμε τις λαθροχειρίες. Έτσι θέλουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να μου απαντήσετε. Αρλίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ ο Πρόεδρος και ευχαριστώ για τις πνευματικέ σου παρατηρήσει όσον αφορά τι προηγούμενε Ιρλανδικέ Προεδρίε. Έχουμε στην προσωπή μας δύο γυναίκε. Είμαστε πάρα πάρα πολύ τρυφεροί και ευγενικοί με τις κυρίες εμείς φοράμε και γραβάτα. Τέλος πάντων, να σας πω τώρα, για να, να σοβαρευτούμε τι γίνεται με το θέμα της ισότητας. Θα πρέπει όντως να θεωρηθεί θέμα προτεραιότητας. Πολύ σοβαρό. Και το παίρνουμε στο σοβαρό. Πρέπει να μιλήσω τώρα σαν Προεδρία, όχι στην Ιρλανδία, αλλά στις εκλογές έχουν ποσοστώσει για τις υποψηφίους. Και ανάλογη είναι και η χρηματοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα. Άρα δεν πρέπει αυτοί να παραβούν τις ποσοστώσεις. Έτσι επομένω θέλουμε να ασχοληθούμε θα σοβαρά τώρα όσον αφορά την οδηγία που αναφέρεται θέλουμε. Αυτό το οποίο προχώρησε από την Υπηρετική Προεδρία να το ολοκληρώσουμε. Για τις κεφαλικές απαιτήσει ε, επίσης το ίδιο και θέλουμε να διευκολύνουμε το έργο του Κοινοβουλίου. Υψίστη προτεραιότητα επομένως. Και αυτό ισχύει για του τρεις πυλώνες. Αν όλα αυτά μπορέσουμε να τα προωθήσουμε στου πρώτους δύο μήνες, τότε ελπίζω ότι πρόκειται να αποκτήσουμε τις επιπλέον πόρου, ώστε να μπορέσουμε ε, όλα αυτά να τα πούμε. Και άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε πρόεδρο για τις οδηγίες αυτές που αναφέρατε κατά το δεύτερο ήμιση της Προεδρίας. Ελπίζω το καταφέρουμε. Κύριε ε, Υπουργέ, αναφέρατε ένα πολύ ε, φιλόδοξο πρόγραμμα, πραγματικά. Ε, αν πετύχετε θα φέρετε την Ευρώπη ένα βήμα πιο μπροστά. Εχθές ο Ολλανδός ε, Υπουργός Οικονομικών ορίστηκε διάδοχος του Ιζάν Πολ Γιούγκερ, αλλά όχι με ομοφωνία, αλλά με πλειοψηφία με σχετικά μεγάλη χώρα, είχε αμφιβολίες. Πώς ε, το αξιολογείτε εγώ, θεωρώ ότι στην αρχή μιας νέας ε, τέτοιας προεδρίας αυτό το αυτή η δυσπιστία ίσως θα μας φέρει δυσκολίες στο μέλλον. Δεύτερον, από την Κύπρο, έρχονται ε, ανησυχητικά μηνύματα. Έχει 8 με 10 εβδομάδες ε, πριν να, είναι, ε, να έχει αφρικιότητα η Κύπρος και υπάρχουν ε, υπάρχει ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία που διοχετεύεται μέσω την Κύπρο και εμείς δεν θα θέλαμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, για το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης αναφέρεται τους τρεις πυλώνες. Ένας από αυτούς τους πυλώνες, ε, το σχέδιο εγγύησης καταθέσεων, έχει εδώ και ένα χρόνο τελειώσει στο Κοινοβούλιο ως θέμα, όμως μόνο ε, μία συνάντηση είχαμε με το Συμβούλιο για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Είστε αισιόδοξοι ότι ταυτόχρονα με την ε, εποπτεία που θα τη συζητήσουμε στις τριμερείς και μαζί με τους άλλους δύο πυλώνες θα μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα μέσα σε έξι μήνες. Και τέλος, όσον αφορά στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, να πω απλώς ε, και να σας ζητήσω να κάνετε κάτι έτσι ώστε στην εσωτερική αγορά να ε, έχουμε ολοκλήρωση εκεί που δεν υπάρχει. Complete the single market, ειδικότερα όσον αφορά στον τομέα των υπηρεσιών. Αν ναι, επιτύχουμε στην ολοκλήρωση το τομέα υπηρεσιών, πραγματικά θα προωθήσουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλίντς. Ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, που ήταν ένας καινούριο στο Eurogroup, έγινε πρόεδρος του Eurogroup εχθές αργά το βράδυ για να διαδεχθεί τον Ζαν Κλοντ γιουγκερ Ο κύριος Μπλουμ είναι πολύ νέος και ταλαντούχος, όμως δεν είναι πολύ γνωστός εντός του Eurogroup. Μπήκε μετά από τις Ολλανδικές εκλογές όταν ε, δημιουργήθηκε η νέα κυβέρνηση. Νομίζω τον Νοέμβρη ήταν η πρώτη του συνεδρίαση, οπότε δεν τον γνωρίζουμε σε προσωπικό επίπεδο πολύ καλά. Παρόλο που έκανε το μάστερ του στο Κόρκ, στην Ιρλανδία. Δεν έχω δει ποιοι ήταν ε, οι βαθμοί του, αλλά ίσως κάποιοι Ιρλανδοί συνάδελφοι να το είδαν. Είναι πολύ ικανός και έχει μια ευρεία άποψη για το τι χρειάζεται να γίνει στην Ευρώπη. Προηγουμένως υπήρχε ένα αίτημα δημόσιο από τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών να μας ε, παρουσιάσει το όραμά του για την Ευρώπη ως πρόεδρος ε, του Eurogroup και το έκανε με μια γραπτή επιστολή σε κάθε μέλος του Eurogroup. Ήταν ο μόνος ε, που διορίστηκε που μάλλον ήταν υποψήφιος παρόλο που είχε ανοίξει ο διαγωνισμός εδώ και μέρες. Φαίνεται όμο, στην αρχή φαινόταν ότι θα είναι ομοφωνή η απόφαση. Τελικά ο Ισπανός πρόεδρος Είχε κάποιε αμφιβολίε, δεν έδωσε του λόγου. Ελπίζουμε όμω ότι θα είναι πολύ καλό ω πρόεδρο και δεν έχω κάποιο λόγο να πιστεύω ότι δεν θα είναι. Τώρα για την κατάσταση στην Κύπρο. Είναι προφανώ σοβαρή. Αν ε, εξετάσουμε το θέμα των Κύπρου με τις τράπεζες και τα κράτη, ε, το όλο ε, ανέρχεται σε 17 και 18, με 18 δις. Είναι ένα μικρό το ποσό σε σχέση με άλλες χώρες. Όμως, αναλογικά με το ΕΠ της Κύπρου, είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει λοιπόν δουλειά για αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν προεδρικές εκλογές ε, στην Κύπρο που περιπλέκουν την κατάσταση και κοινοβουλευτικές εκλογές έτσι λοιπόν οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν την κατάσταση της Κύπρου και η παρούσα κυβέρνηση στην Κύπρο έχει θεσπίσει μια σειρά μέτρων που θα απαιτηθούν αν μπει στο, αν μπει στο πρόγραμμα η Κύπρος Περιμένουμε λιγάκι. Δεν θα έχουμε καταλήξει πριν τις εκλογές μάλλον στην Κύπρο, αλλά όπως και να έχει θα είναι ικανοποιητικό θεωρώ το αποτέλεσμα για την Τραπεζική Ένωση. Η αλληλουχία έχει ως εξή. Ο ενιαίος ο μηχανισμός εποπτείας πρέπει να ολοκληρωθεί στην τριμερή και μετά να ε, δημοσιευθεί το έγγραφο του ψηφίσματος και η ε, οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις 4 πρέπει να εφαρμοστεί και τότε θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που έρχονται. Η εγγύηση καταθέσεων θα πάει ταυτόχρονα με τη διαδικασία ανάκαψης και εξυγίανσης. Η αρχική πρόταση ήταν να έχουμε ένα μείγμα των εθνικών συστημάτων εγγύησης, όμως ε, το χρονοδιάγραμμα μάλλον μας πιέζει. Αλλά θα έχουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Ναι, η σταθερότητα, η θέση εργασίας και η ανάπτυξη είναι τα θέματα της Προεδρίας μας σε χώρες ε, που βρίσκονται σε δύσκολες ελληματικές θέσεις. Με έλλειψη πόρων είναι δύσκολο να έχουμε ένα πακέτο ή, τύπου New Deal. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά. Δεν είναι ευθύνη του ΕΚΟΦΗΝ, όμως σε επίπεδο υπηρεσιών και ειδικά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική η ολοκλήρωση της αγοράς. Είναι μόνο 80% ολοκληρωμένη η αγορά και φυσικά θα υπάρχει σημαντική απόδοση σε επίπεδο ε, θέσπισης θέσεων εργασίας αν υπάρξει ολοκλήρωση και γι' αυτό θα είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Ωραία. Περνάμε τα πέντε λεπτά γιατί είναι και μεγάλες και ερωτήσεις για το ECR Σαέτ Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ Γιατί ένα από αυτά τα θέματα που θα σα πω είναι τα θέματα τα οποία μα απασχολούν, το θέμα για την ομοθεσία δηλαδή το τι θα κάνουμε με τα τράπεζε που χρεοκοπούν και μετά θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να τη στηρίξουν. Γιατί έχουμε τρία τιμά που θα θέλαμε εμεί η ΙΣΙΑ να δούμε. Επομένω, να μην γίνεται διάσωση βάρος λοιπόν να αποδέονται ευθύνε σε αυτού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και να μην φέρουν ευθύνη μόνο να πληρώνουν την ύφη οι φορολογούμενοι και επίση να υπάρχουν κάποια, κάποια στάνταρ τόσο ώστε να έχουμε σωστή καταγραφή, λογιστική καταγραφή των ζημιών και θα πρέπει να δούμε το ότι στις καλές εποχές επομένως καρπώνονται τις, τα κέρδη και μετά πρέπει άλλος να στηρίξει και να πληρώσει για τις ζημίες μετά. Άλλωστε έτσι καταστράφηκε η δική σας οικονομία. Όταν είχε πραγματικές ζημίες με το πραγματικές οικονομίες η κάθε σας τράπεζα. έχουμε την οδηγία, τη συμφωνία IFRS για τις τράπεζες και θα έπρεπε να ε, συμμορφώνει οι τράπεζε. Επίση. τι λέτε, πώ αυτό το IFRS θα καταστεί συμβατό με το, με με το Βρετανικό δίκαιο και ειδικά με τα όσα διέπουν τη λογιστική. Σας ευχαριστώ κύριε Καμάλ. Αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά την κατανομή του, του βάρους και τη ζημία με του φορολογουμένου. σε σχέση με τη διάσωση, σε σχέση με το δεν έχουμε κάποια στάνταρ λογιστικής. Και επομένως θα πρέπει να το δούμε. Τα άλλα τα οποία είπατε. αφορούν περισσότερο την ιδιωτά μου Ιρλανδού Υπουργού. Έχετε δίκιο. Ήταν απαράδεκτη η κακοδιαχείριση που γινόταν. Υπήρχε αυτή η παράδοση ούτως επίνου της επίοικούς εποπτείας επί των τραπεζών και το σύστημα δούλευε επί τη βάση κάποιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης που τελικά ήταν αβάσιμη, δικαιολόγητη έχουμε τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης που είδαμε τι κάνανε στην Αμερική γιατί είχαμε εκείνα τα ομόλογα τα οποία κατέληγαν να είναι σκουπίδια παρά τις αξιολογήσεις που του. Άρα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν και ο φορολογούμενος. Στην Ιρλανδία προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να επαναρθώσουμε τη ζημία που έγινε και επίση να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να σα πω τόσο πολλά και εμεί ένα βιβλίο, αλλά δεν θα τα πω και θα βάλω τελεία εδώ. Και σα ευχαριστώ, Πρόεδρο. Θέλετε να δευτερολογήσετε, γιατί έχετε ακόμα χρόνο. Καμάλ, ναι. Γιατί ε, αυτό που ρώτησε στο τέλο όσον αφορά του οικονομικού ελέγχου, του IFRS, αυτό, αυτό δεν, δεν αφορούσε την Ιρλανδία. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς από πολλές χώρες. Έχουν έρθει και μου έχουν βρει πολλοί και μου έχουν θέσει το πρόβλημα. Τεχνικό θέμα αυτό. Αλλά εγώ σας είπα τι θα κάνετε σχέση με την Κομισιόν που, που τις έχουμε ζητήσει να αναθεωρήσει το IFRS ε, το, το, για να είναι συμβατός με το δικό μας δίκαιο αυτό γιατί για τη διαχείριση των εναλλακτικών επενδύσεων δηλαδή. Δεν είναι θέμα το ΕΚΟΦΗΝ όμως, λέει ο Υπουργός. Θα συζητηθεί αναθεώρηση του κειμένου σε άλλο συμβούλιο. Και ο Ρίτσαρντ Μπρούτον, υπουργό τον έχει απασχολήσει το θέμα, το αυτό συζητήθηκε σήμερα εδώ στην ΙΜΚΟ, στο Κοινοβούλιο. Για την εποπτεία. Δεν έχει υποθεί ακόμα τίποτα επίσημο. Γι' αυτό και προβληματιζόμαστε τι θα γίνει. Όχι ο Σβέν, αλλά ο Φιλίπιος Κωσίνης. Σας ε, καλωσορίζω στην πόλη μου της Βρυξέλλες, κύριε Υπουργέ. Από την έναρξη της Ιρλανδικής ε, Προεδρίας α, μας είπατε πολλά καλά λόγια. Σας πιστεύουμε, σας πιστεύσαμε μέχρι να μπούμε σε διαπραγματεύσει. Μιλάω για δύο θέματα, το SSM που είναι στο εκοφήν και το άλλο είναι το, η Βασιλεία 3 που λέγεται και αλλιώς ε, απατήσεις ή σχετική οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων νούμερο 4. Ποια είναι η στάση σας. Ο, λέτε ότι η, ο συμβασμός στο Συμβούλιο ήταν τόσο δύσκολος να επιτευχθεί που δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε. Αυτή ήταν η στάση σας. Για την τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, το μήνυμα ήταν, ήταν περίπλοκο το θέμα, μεγάλο το θέμα και ό,τι κι αν πιστεύετε, ε, ακόμα και αν πιστεύετε ότι συμφωνείτε, ε, κάνετε λάθος, εμείς θα το ξανανοίξουμε το θέμα, ό,τι κι αν συμφωνήθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας, εμείς θα το ξανανοίξουμε. Βέβαια, το είπατε πιο διπλωματικά από τα λέω, δεν μπορώ να τα πω το ίδιο όπω τα είπατε. Αν όμω αυτή είναι η στάση του Συμβουλίου, δηλαδή τη στιγμή ε, τα στυλώνει και στην άλλη καθυστερεί, δεν νομίζω ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Για το CRT, στέλνετε διπλωμάτες, αλλά κάποια στιγμή ε, τα θέματα αυτά είναι, θα δείτε ότι είναι πολύ πολιτικά, ε, με υψηλό τίμημα, σας θέλουμε εκεί για να κλείσουν αυτά τα σημεία. Γιατί δεν μας αρέσει το Συμβούλιο να θεωρεί ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των τραπεζών χωρίς να ε, ετοιμάζεται να πει κάποια πράγματα, μπορεί να πει κάποια πράγματα ανοιχτά και να είναι και σε θέση να πληρώσει και το πολιτικό τίμημα. Λυπάμαι που είναι αυτή η εντύπωση σας κύριε Λάμπερτς για την τέταρτη ε, ε, οδηγία για τις κεφαλαίκες απαιτήσει το αποτέλεσμα οποιοδήποτε τριλόγου θα πρέπει η συνεχεία να εγκριθεί από τα 26 κράτη-μέλη. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Και οποιαδήποτε απόκληση από τη θέση του Συμβουλίου πρέπει να συμφωνηθεί ομόφωνα στο ΕΚΟΦΗΝ. Τον περασμένο Μάιο ε, συζητήσαμε και συμφωνήσαμε σε υπουργικό ε, επίπεδο. Μέχρι να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία πραγματική. Θέλουμε να συμφωνήσουμε, ε, δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε το κείμενο, θέλουμε να το ενοποιήσουμε, να το παγιώσουμε. Θέλουμε να συμφωνήσουμε γρήγορα και μάλιστα νωρίς την Προεδρία μας. Για το SSM επικρίνεται πάλι τις ε, διαπραγματεύσεις μας. Εγώ νομίζω ότι προχωράνε τα πράγματα και έχει σημειωθεί πρόοδο. Το SSM που είναι ο ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Αυτό περίμενα να μου πείτε, κύριε Υπουργέ, λέει ο κύριο Λάμπερτ. Αλλά για το SSM χρειάζεται ομοφωνία. Αλλά για κάποια τμήματα του φακέλου χρειάζεται και το κοινοβούλιο. Για το CRD, για τι κεφαλαίκε απαιτήσει, δεν χρειάζεται 26 κράτη-μέλη μαζί σα, μαζί με την Προεδρία. Από ό,τι ξέρω, δεν ε, λαμβάνεται εκεί ε, απόφαση ομόφωνα στο Συμβούλιο. Εάν σας λένε ότι η διαφάνεια ή η περιστολή των υπερβολικών πόνους ε, του κλάδου δεν θα πρέπει να είναι τμήμα του, της νομοθεσίας αυτής, τότε θα έρθουμε σε αντιπαράθεση, τότε θα υπάρξει διελκυστίνδα μεταξύ ημών και θα λάβει και δημόσιες διαστάσεις. Ξέρω ότι αυτά που λέτε είναι θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Ο ρόλος μας είναι να διευκολύνουμε τη συμφωνία, λέει ο υπουργό. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε την Ιρλανδική άποψη στο Συμβούλιο. Για την τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαίκες απαιτήσει, η αρχική μας προσέγγιση είναι να παγιώσουμε αυτά που συμφωνήθηκαν όταν έχουμε αυτό το συμπεφωνημένο κείμενο, μετά μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπήρχαν όμως κάποιες αμφισημίες για κάποια από τα θέματα. Θέλουμε να προχωρήσουμε με βεβαιότητα. Θα πρέπει να έχουμε σίγουρα κάποια δεδομένα, ας πούμε, όλο το κείμενο και μετά να προχωρήσουμε. Η Μαρίσα από την Γκουε. Ευχαριστώ. Καλώς σας καλωσορίζω κύριε Υπουργέ. Θέλω να μιλήσω για κάποια αποτελέσματα του ΕΚΟΦΗΝ. Να μπω σε λεπτομέρειες όμως. για τη δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας των δανείων. Ε, μέρους του χρέους της Ιρλανδίας. Αυτό δεν συνδέεται όμως μόνο με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και με το μηχανισμό στήριξης. Αν το χρέος σας ε, είναι μη βιώσιμο, πώς γίνεται αυτό. Ακόμα και αν ε, επιμικίνουμε τη διάρκεια αποπληρωμής του χρέους, δεν λύνεται το πρόβλημά σας. Επίσης, τι ελπίζει να πετύχει ως συμφωνία η Ιρλανδική κυβέρνηση για τα γραμμάτια, ε, είναι ένα θέμα που τέθηκε. Ποια θα ήταν για σας μια καλή συμφωνία για τα γραμμάτια. Ε, thank you very much indeed, ε, Ευχαριστώ κυρία Ματίας, λέει ο Υπουργός, για το Eurogroup και την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών της Πορτογαλίας. Η Κομισιόν είπε ότι θα αποτανθεί σε, σε μια ομάδα ανώτατων υπαλλήλων για να δουν τη δυνατότητα κατά πόσο μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων ε, δανείων Ιρλανδίας και Πορτογαλίας. Ιδίως ε, τα δάνεια που ε, έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για το EFSM, e εκεί όμως η απόφαση για τα δάνεια από το EFSM ε, λαμβάνονται ε, και από τους 27 και όχι από το Eurogroup. Που είναι ο μηχανισμός σταθερότητας. Ε, στη μία περίπτωση αποφασίζει το Eurogroup, στην άλλη περίπτωση αποφασίζει το ECOFIN. Ο Βιτόρ Γκασπάρ, ο Πορτογάλος υπουργό μίλησε ξανά και είπε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση στο ECOFIN με την στάση του Eurogroup. Η συμφωνία ήταν ότι υπό την ευθύνη της Κομισιόν ανώτατοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι θα εξετάσουν τη δυνατότητα για την οποία ζητήσαμε και θα μας ενημερώσουν στη συνάντηση του Μαρτίου. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, για τα κραμάτια, οι σχετικές διευθετήσεις προβλέφθηκαν για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων αφαιρέγγιων τραπεζών. Ε, οι τράπεζες μας φτάσαν σε αφαιρεγγιότητα ε, μετά από προβλήματα με τις ε, κατασκευαστικές εταιρείες. Πήραμε δάνειο και η αποπληρωμή αυτών των δανείων ήταν πολύ μικρή, μικρή προθεσμία. Επιδεινώνεται η κατάσταση από το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση συμφώνησε για τα επιτόκια. Ε, επιτόκια πολύ ψηλά. Είπαμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή, είπαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε αυτά τα γραμμάτια και θέλουμε μεγαλύτερες ε, διάρκειες αποπληρωμής και χαμηλότερα επιτόκια. Συμφωνήσαμε επί κάποιων σημαντικών θεμάτων, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και στις δύο διαπραγματεύσεις υπάρχει και το θέμα της διαγραφής των δανείων ε, και της πτώχευσης. Ε, αλλά αυτό δεν, το θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμεί θέλουμε απλώ μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμή και χαμηλότερα επιτόκια. Ούτω ώστε να είναι πιο βιώσιμα τα κρατικά χρέη. Να έχουν αυτή τη δυνατότητα τα κράτη, ούτω ώστε να έχουν πιο ε, εύκολη πρόσβαση στι αγορέ ομολόγων. Ο Πίτερ Μάρτιν. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ανησυχία που πολλοί από όσους ε, χαράσουν πολιτική και πολλοί πολίτες έχουν. Έχουμε την εντύπωση ότι στην Ιρλανδική Προεδρία υποστηρίζεται κάποιες θέσεις που ήδη έχει επιτύχει η Κυπριακή Προεδρία. Θα ήταν λάθος πίνημα ε, μέσα από τις ε, εμπειρίες που είχατε εσείς με την έλλειψη ελέγχου στις τράπεζες ε, και το βάρος στους φορολογούμενους, τώρα να πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα μια ερώτηση για την έκθεση Λικάνεν. Ποια είναι η άποψή σας για τις προτάσεις που έχουν γίνει. Θεωρείτε ότι είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να υποστηρίξει η Ιρλανδική Προεδρία και αν ναι, τι θα πιστεύετε για την ανακοίνωση του κυρίου Μπαρνιέ να υπάρχει πρόταση μέσα στην Προεδρία σας θα το επιδιώξετε ή θα πείτε ότι δεν σας αφορά. Uh, είναι άδικο να πούμε ότι κάνουμε πίσω τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Είχαμε τρεις τριμερείς ήδη και για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις τέσσερα είχαμε δύο. Ήδη ε, από την 1η Ιανουαρίου έχουμε την Προεδρία, σήμερα είναι 23 Ιανουαρίου και έχουμε δώσει κατάλληλη προσοχή και στα δύο θέματα. Τρεις τριμερείς στη μία περίπτωση και δύο στην άλλη. Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε διαμεσολαβητές για συμφωνία όχι να επιβάλλουμε τις Ιρλανδικές απόψεις. Δεν υποχωρούμε σε καμία περίπτωση και ούτε θέλουμε να κάνουμε πίσω. Όπως είπα πριν, για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις 4 υπάρχει διαφορά απόψεων με, σε αυτούς ε, με τους οποίους ε, ερχόμαστε σε επαφή με βάση τα, πόσα, τα όσα συμφωνήθηκαν και προσπαθούμε να βασιστούμε στα όσα συμφωνήθηκαν για να πάει μπροστά το ψήφισμα. Για τις προτάσεις Ελικάνεν, περιμένουμε πρόταση, ε, όμως μάλλον δεν θα προταθεί αυτή πριν το πέρας της Προεδρίας μας, οπότε να έρθει, θα έρθει μάλλον Μάιο-Ιούνιο και δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε εμείς να ασχοληθούμε θέλετε να επανέλθεις, Πίτερ. Μια επιπλέον παρατήρηση για τον συνάδελφο Φίλιπ Λάμπερτς. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν γίνονται οι συναντήσεις, αλλά ότι υπάρχουν διπλωμάτες και η άλλη πλευρά ακούει ότι ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Και αυτό καλό θα ήταν να το έχετε στο μυαλό σας ως υπόβαθρο για να γνωρίζετε ποια είναι η αντίληψη που υπάρχει στο Κοινοβούλιο και σε όσους ε, βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση. Το να έχεις διπλωμάτες και ανώτατους αξιωματούχους ε, ε, είναι μια στάνταρ διαδικασία όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπουργοί είναι από τις κυβερνήσεις που δίνουν τις ε, οδηγίες και οι οδηγίες είναι να επιληθούν τα θέματα αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί δεν έχει γίνει ε, καμία πρόοδος. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε ότι έχουμε διάφορα θέματα σε διάφορα στάδια προώθησης, ε, ε, η επιτυχημένη Προεδρία είναι αυτή που έχει ολοκληρώσει θέματα. Και εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσουμε ε, με τη σειρά που ανέφερα στην αρχική μου παρουσίαση τα θέματα που παρουσίασα. Και θέλουμε να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και τις θέσεις του Συμβουλίου ταυτόχρονα. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας διακόψω για να σας πω ότι η Ελληνική Προεδρία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί από το, από το χρόνο που τους έχουμε δώσει, αλλά δεν θα τους αφήσω γιατί θα πρέπει να, να, να, να, ελέγξουμε τη, τη συνεδρία. Ε, πρόεδρος, με τι να κάνουμε. Γκέι Μίτσελ. Γκέι Μίτσελ, για το ΕΛΚ. Σας γνωρίζω, κύριε νιούναν πολλά χρόνια. Και ό,τι, όσο και να, και, και να σας κάνω κομπλιμέντα, θα δώσουν εντύπωση ότι κολακεύω. Νομίζω ότι αυτά τα οποία κάνετε πάντως ήδη μέχρι τώρα για την ανάκαμψη της χώρας νομίζω ότι ήταν υποδειγματικό. Και ήταν ο Μπρένταν Μπίχαν, ξέρετε, ένας ε, θεατρικός συγγραφέας. Ξέρετε τι είχε πει αν κανένας έχει, έχει, έχει ψάρια μπορεί να κάνει fish and chips, αλλά μόνο με πατάτες. Αυτό αφορά και αυτό το οποίο έχετε πετύχει. Νομίζω ότι θα πρέπει την ε, επιτυχία να την πιστωθεί. Ο δημόσιος τομέας για τη συνήθως επικρίνεται και εδώ και αλλού. Όταν λαμβάνονται όμως από το κράτος κάποιες σκληρές αποφάσεις, θα πρέπει όλοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Και Έχει ρίξει μια τέτοια και στη ΣΥΠΑ. Υπουργέ, για πετε μας. Έχετε κάποιες ενδείξεις για το ότι τελικά θα σταματήσει η κερδοσκοπία κατά του ευρώ, κατά των αγορών, κατά της Ευρώπης. Και η Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει το ευρώ. Εγώ θέλω να τονωθεί η επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει να μην τζογάρουν οι επιχειρηματίες, θα πρέπει να διακινδυνεύουν ελελογισμένα. Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει η Κεντρική Τράπεζα, γιατί τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν ε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή φέτος. Τέτοια μέτρα θέλει ο κόσμος. Τι θα γίνει, τι λέτε. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Προβληματίζει πολύ αυτό το οποίο ρώτησες. θα πρέπει κανείς να εξετάζει τι έχει συμβεί στο παρελθόν για να σχεδιάσει το μέλλον. Ένα σωρό πολιτικές είχαμε, μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Τη διπλή δέσμη, την εξαπλή δέσμη, το σύμφωνο σταθερότητας, τα διάφορα ταμεία, το μηχανισμό σταθερότητας, κλπ. Είχε γίνει πρόοδος, σίγουρα. Σκεφτείτε πώς ήταν η Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2012 και, και, και πώς είναι τώρα η Ευρώπη το 2013. Πολύ σταθερότερη τώρα. Άρα αποδίδουν τα όσα έγιναν. Και βέβαια θα πρέπει να πάρει συγχαρητήρια και η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα. Βοήθησε πολύ. Νομίζω ότι το ρίσκο και κίνδυνο κάθε φορά αντικατοτρίζονται στα επιτόκια. Τα επιτόκια είναι ψηλά ή χαμηλά, ενώ είναι ψηλός ή χαμηλός ο κίνδυνος. Σε εμά η τάση χαμηλο ο κινδυνο σε εμα πτωτική. Το ίδιο και για το μηχανισμό στήριξη. Αυτό ενθάρρυνει τους επενδύτες. Ούτε ισχύει όμως ότι κερδίσαμε το παιχνίδι και πια δεν έχουν προβλήματα. Ακόμα συνεχίζεται η πορεία μας. τελικά αυτό μετράει είναι το κατά πόσο καταστρέφεται ο κόσμος. Γιατί η ανεργία είναι τρομερή στην Ευρώπη. Και η ανεργία των νέων. Απαράδεκτα επίπεδα για δημοκρατικές χώρες. Αλλά θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Αυτό θέλει να κάνει η Προεδρία μας. Όλα αυτά θέλουμε όχι μόνο να μας ασχολούν εμάς, αλλά θέλουμε και να, να είναι η βασική άξονα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για αυτό το εξάμεινο. Και κάπως έτσι να βοηθήσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ελκ, πάλι. Γιώργο. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον Υπουργό και θέλω να του πω ότι έχω μεγάλες προσδοκίες από την Προεδρία του. Στο παρελθόν είδαμε Ιρλανδικές Προεδρίες τρομερές, πολύ επαγγελματικές, πολύ αποτελεσματικές. Πιο πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, στο εσωτερικό της Επιτροπής μας, είχαμε υποδεχθεί τον ε, κύριο Γιούνκερ και μας είπε ότι χωρίς αυτόν τα κράτη που είναι υπομνημόνιοι υπό πρόγραμμα τέλο πάντων και που έχουν συμφωνία με την Τρόικα, χωρίς αυτόν, ε, ή μάλλον είπε ότι αυτά τα κράτη μπορούν να πάρουν κάποια χρήματα. Κάποια αποζημίωση, μας είπε για ποια αποζημίωση, για ποια χρήματα μιλάμε ε, για αυτά τα κράτη που έχουν αυτά τα μνημόνια ή αυτά τα προγράμματα. Uh, Σίγουρα οι χώρες και οι πληθυσμοί βρίσκουν δυσ... πολλές δυσκολίες να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Τους τελευταίους 12 μήνες όταν ανοίγουμε τις ε, βραδινές ειδήσει, βλέπουμε πόσες κοινωνικές αναταραχές υπάρχουν, πόσες διαδηλώσεις στους δρόμους. Στις χώρες ε, υποδιάσωση, ε, οικογένειες, άτομα περνάνε πολύ δύσκολα. Τα επίπεδα ανεργίας είναι πολύ ψηλά, οι υπηρεσίες είναι πολύ χειρότερες, ας πούμε στην παιδεία, ε, αυξάνεται, είναι χειρότερες οι υπηρεσίες, ε, αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης, ε, το άμεσο εισόδημα μειώνεται, μειώνεται το βιωτικό επίπεδο επίσης. Αν αυτό διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυσικά η ευημερία θα πληγεί. Ω πολιτικοί δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις δυσκολίε που έχουν ορισμένε χώρε, ειδικά οι χώρε ε, υποδιάσωση. Θα πρέπει να τίνουμε χείρα προς τους νέους ειδικά, γιατί με αυτά τα επίπεδα ανεργίας που τους πλήττουν, ειδικά σε ορισμένες χώρες, η κατάσταση είναι αβίωτη. Δεν είναι δυνατόν δημοκρατικές χώρες να έχουν τέτοια υψηλά επίπεδα ανεργίας. Κάτι πρέπει να γίνει. Σε ό,τι αφορά τα πακέτα αποζημίωσης. Διάφορες προτάσεις έχουν ακουστεί για να διασκεδάσουν τις δυσκολίες των κρατών μελών. Αλλά για το πώς θα καταστεί το χρέος πιο βιώσιμο και πώς θα επιμηκυνθεί η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων, εκεί χρειάζεται έχηση χρήματος. Ξέρετε, ένα κυρίαρχο κράτος, ας πούμε, ξέρει τι πρέπει να δαπανίσει για να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Η λύση είναι να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ανάπτυξη οδηγεί στην εξέβρεση λύσεων. Η λιτότητα δεν βοηθάει σε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε στρατηγικές για ανάπτυξη, για θέσεις απασχόλησης. Είναι εκ των όνων κάνευ αυτό. Αυτό το αναγνωρίζουμε πια. Το αναγνωρίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές, το αναγνωρίζουν και οι αρχές των κρατών μελών από το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μπράβο για αυτά που είπατε για τους νέους στην ανεργία και για το ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί αυτή η τρομερή κατάσταση. Υπάρχει κι άλλος θεατρικός συγγραφέας που ο Γκέι Μίτσελ δεν τον θυμήθηκε. Τον Όσκαρ Βάιλ. Ναι. Και εκείνος έλεγε ότι οι φιλοδοξίες είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Και πολύ καλό να τα λέμε, να τα σχεδιάζουμε, αλλά θα πρέπει κάπως να δούμε ότι μέτρα, τα μέτρα και οι δεσμεύσεις είναι κάτι το οποίο ε, καταραίει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε για πετε μας. Πιο συγκεκριμένα, τι θα κάνετε κατά την Προεδρία σας. Ο Ντάισελμπλουμ, ο Υπουργό Οικονομικών μας, θεώρησε ότι τώρα έχει ανανεωθεί η εμπιστοσύνη προς το ευρώ, οπότε μπορούμε να φροντίσουμε την ανάπτυξη. Άρα, μήπως θα πρέπει να συνεργαστείτε με το Eurogroup. Να αποφύγουμε τον διχασμό μεταξύ αυτών που είναι μέσα και αυτών που είναι εκτός Eurogroup. Υπάρχει αυτή η δεσμή μέτρων για την ελληνική των Νέων και για του αμέσω επόμενου μήνε πρόκειται αυτό να ζητηθεί από του υπουργού. Δεν έχω υπόψη μου το πιο συγκεκριμένο, αλλά θεωρώ ότι οι λεπτομέρειε του θέματο είναι γνωστέ. Εκπαίδευση, περισσότερη κατάρτιση για τους νέους. Να προσέχουμε πού πάνε για να πιάσουν δουλειά, για να αποκτούν κάποια εμπειρία. Και φυσικά μέτρα ανάλογα με κάθε συγκεκριμένη χώρα. Βεβαίω και ο κύριος Ντάσελμπλουμ θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και θα συνεργαστούμε μαζί. Τώρα όσον αφορά την ιδέα για την εγγύηση για την απασχόληση των νέων. Θα το προωθήσουμε αυτό. Αυτό υπάρχει σε τα δεκαετία του 70 στην Ορβηγία και αποδίδει. Δεν έχουν στην Ορβηγία ιδιαίτερη ανεργία στους νέους. Ίσα ίσα να απασχολούν και Σουηδούς, νέους Σουηδούς. Επομένως αυτό θα μας απασχολήσει εντόνως. Πρόεδρος, θέλετε να ρωτήσετε κάτι Ναι, ναι, ζήτησα κάτι για την ε, διαίρεση, για το διχασμό μεταξύ των εντός και των εκτός Eurogroup. Το νόμισμα διχάζει. Άλλοι το έχουν, άλλοι δεν το έχουν, αλλά 27 θα πρέπει όσο γίνεται να συνεργαστούν. Να συνεργαστούν για μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα, όπως ας πούμε η ενεργεία των νέων. Αυτό είναι κοινό θέμα, ό,τι και να ισχύει νομισματικά σε κάθε χώρα. θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σωστή πολιτική είναι αυτή που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Άλλοι τρεις θα λάβουν το λόγο. Ο Γκούνε, η Άννη Ποδηματά και συνέχεια και άλλοι. Ευχαριστώ. Κάποια από τα σημεία και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε είναι διαφορετικά σε χαρακτήρα από άλλα. Κάποια ε, είναι στον ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και είναι σχεδιασμένα για όλη την Ένωση, ενώ άλλα είναι σημεία που συζητούμε μέσα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω από εσά την άποψή σας για τους κινδύνους. Βλέπουμε κάποια φυγόκεντρες δυνάμεις εδώ. Έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Αυτό είναι κομμάτι των μελλοντικών ε, δυνατοτήτων. Όμως ο, ο κίνδυνος είναι ότι δημιουργούμε δομές οι οποίες πιο πολύ διχάζουν παρά ενώνουν. Για παράδειγμα, πολύ συχνά μιλάμε για τους ε, μέσα και τους έξω. Αυτούς που είναι στην Ευρωζώνη ή όχι, αυτοί που επιλέγουν να είναι μέσα ή όχι, βοράς, νότος. Αναρωτιέμαι, πώς εσείς βλέπετε τη δική σας ευθύνη, τη δική σας δυνατότητα να διασφαλίσετε την Ενωμένη ε, Ένωση. Να πω, να πω και σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες ε, για την οδηγία εξηγήνσης και ανάκαμψης. Επειδή είμαι ο εισηγητής, θα ήθελα να ακούσω πού είναι τα πολλά προβλήματα στο Συμβούλιο. Γιατί όπως είπατε πριν, το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ αισιόδοξο, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον. Το να τελειώσει δηλαδή αυτό το θέμα στην Προεδρία σας. Καλό θα ήταν, αλλά αυτό σημαίνει ότι από νωρί θα πρέπει να ορίσουμε τα βασικά προβλήματα για να τα λύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Ευχαριστώ. Κύριε Χοκμάρκ, για την πρώτη σας ερώτηση σχετίζεται σε επίπεδο αρχής με την ε, συνοχή της Ένωσης. Αναφέρατε τον Βορρά και τον Νότο και, άλλες τέτοιες, και διαχωρισμούς. Ένα από τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι ότι εδώ και τώρα μερικά χρόνια επικεντρωνόμαστε πλήρως στα ελλείμματα και στους ισολογισμούς ενώ η πραγματική έγκλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πιο ουσιώδης και πιο ιδεαλιστική. Η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η δημοκρατία, των ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν οι χώρες της πρώην Σοβιετικής ε, Αυτοκρατορίας ε, είδαν ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ελκυστική για αυτούς, ε, το είδαν γιατί είχε κάποιες πολιτικές ε, η Ευρώπη και κάποιες θεμελιώδεις αρχές δημοκρατικές. Αυτές οι δημοκρατικές χώρες που είναι αφοσιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα εξυπηρετούν τους πολίτες τους, τους καθιστούν ικανούς να ζήσουν μια ε, ζωή μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και αυτό αρέσει σε αυτές τις χώρες, όπως και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, που κοιτάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν ελκυστικό τόπο εργασίας και διαβίωσης. Κάποιοι από τους ε, ηγέτες σας ε, που έχουν παγκόσμια εμβέλεια δείχνουν ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μόνο τα ελλείμματα που μας απασχολούν. Ουσιαστικά συνάδουμε με τις ε, ιδέες των ε, πατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι η συνοχή ε, είναι ένα από τα θέματα του ΕΚΟΦΗΝ και των Υπουργών Οικονομικών. Τώρα για την ε, οδηγία για την εξηγένση. Αντιμονούμε να συνεργαστούμε επί της οδηγίας για τις τράπεζες. Θεωρούμε ότι είναι πολύ φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα. Θα προσπαθήσουμε όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σκληρά να επιτύχουμε τους στόχους που που θέλετε. Τα βασικά θέματα δεν διχάζουν τόσο, επί της αρχής τουλάχιστον. Αλλά η αλληλουχία και η αναλογικότητα, οι εθνικές, ε, η εθνική διάσταση είναι πράγματα που μπορεί να, καθυστερήσουν, να μας καθυστερήσουν, αλλά υπάρχει καλή θέληση. Παρόλο που είναι στενό το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Έχω άλλους τρεις. Άννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω, Υπουργέ, και σας εύχομαι επιτυχία για την Προεδρία σας. Ξεκίνησε εγώ νομίζω καλά, γιατί στο πρώτο ΕΚΟΦΗΝ που προεδρεύσατε σήμερα υιοθετήσατε την απόφαση για την έγκριση σε 11 κράτη-μέλη να προβούν στην επιβολή φόρου χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Τώρα περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν σχετικά. Ξέρετε άραγε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την διαδικασία λήψη των αποφάσεων στο Συμβούλιο και αν εσείς θα λάβετε περαιτέρω δράση ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας επί του θέματος αυτού για τη φορολογία πάντα, που είναι μία από τις προτεραιότητές σας κάτι που βρίσκω πολύ θετικό. Θα ξέρετε ότι εν ώψη της 50 επαιτίου της ε, συνθήκης των Εκκλησίων, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ηγέτες είπαν χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ε, συντονισμό των φορολογικών πολιτικών και εναρμόνιση των φορολογικών καθεστώτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Και να μειώσουμε επίσης το φορολογικό ανταγωνισμό και το φορολογικό dumping. Ποιες είναι οι απόψεις σας από ε, αυτού του θέματος. Σκοπεύετε να λάβετε κάποια δράση επί των θεμάτων αυτών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ κύριε Ποδηματά. Για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τα επόμενα βήματα είναι ότι η Κομισιόν θα υποβάλει ένα έγγραφο που θα καθορίζει με ουσιαστικό τρόπο τα στοιχεία που θα αποτελούν αυτό το φόρο και η Ιρλανδική Προεδρία θα προεδρεύσει των συνεδριάσεων όπου θα συζητηθεί αυτός ο φόρος και εμείς θα παίξουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή. Όσοι διαφωνούν με, το, με την επιβολή αυτού του φόρου, φυσικά θα συμμετάσχουν πλήρως. Δεν πρόκειται να γίνει διάλογος μεταξύ των 11 κρατών που επέλεξαν την ενισχυμένη συνεργασία. Όλοι θα εμπλακούν και εμείς θα παίξουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή για να υπάρξει προώθηση του θέματος. Για την φορολογική εναρμόνιση αυτό είναι ένα επιπλέον βήμα. Προς το παρόν έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε το πρόγραμμα του Επιτρόπου Σεμέτας για να καταστήλουμε την φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους και θα προωθήσουμε το πρόγραμμά του και θα συνεργαστούμε πλήρως μαζί του. Ο Λίαμ. Εσύ και μετά θα έχω και άλλες δύο ερωτήσεις που θα τις, βάλω, θα τις ακούσουμε μαζί. Ο Λίαμ. Ευχαριστώ, Σάρων. Συγγνώμη που ε, καθυστέρησα. Ήμουν σε μία ε, συνεδρία με τον Μάρκο Μπούτη από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ. Ε, θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα που του έθεσα. Γιατί μιλούσαμε για την σημερινή έτσι, κακή συγκυρία που θα ζήσει και η Ευρώπη το 2013. Το Six Pack προβλέπει ένα ρυθμό μείωσης των ελλημάτων 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο και ο ρυθμός που επιβάλλει η Κομισιόν είναι 1,5%. 1,5% του ΑΕΠ μείωση των ε, ελλημάτων. Όλοι ξέρουν ότι περισσότερες χώρες δεν θα τα καταφέρουν το 2013. Θα γίνει σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο, ούτως ώστε οι χώρες που το ζητούσαν και το πέτυχαν να μπορέσουν να μειώσουν ε, το έλλειμμά τους με βάση το προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα, ούτως ώστε να παίξουν οι αυτόματοι σταθεροποιητέ. Επίσης, η Κομισιόν δημοσίευσε ένα προσχέδιο, ένα blueprint, που επαναφέρει προτάσεις που και ο κύριος Φανδρόπου θα μπορούσε να αναπτύξει στο έγγραφο που θα υποβάλει. Και λέει ότι στην Ευρωζώνη δεν μπορεί να λειτουργήσει το πράγμα χωρίς προϋπολογισμό για να διαχειριστούμε τα ασύμετρα σοκ, δηλαδή τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ε, δυσκολευόμαστε να πληροφορηθούμε για τη συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Έθεσα το θέμα στον κύριο Γιούνκερ. Πώς θα ε, τροφοδοτήσετε τους ίδιους πόρους αυτού του προπολογισμού της Ευρωζώνης. Ε, μήπως ξέρετε κάτι παραπάνω από εμά. Και εν συνεχεία ο Αντολίν θα σας θέσει και αυτός ερωτήσεις γιατί αποφασίσαμε να μοιράσουμε το χρόνο μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία γιατί έταξε ως προτεραιότητα την οδηγία για τα στεγαστικά. Αυτό είναι επίδειξη ρεαλισμού και για μας πάντως είναι μια προτεραιότητα. Και με αυτό το ρεαλισμό ελπίζουμε τελικά να μπορέσουμε να, να προβούμε σε κάποιο είδου σημαντικέ δεσμεύσει, ούτω ώστε να βγάλουμε ει πέραν την εντολή που είχε αναλάβει η Επιτροπή μα. Οπότε και ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επόμενη, ε, στην επόμενη φάση, ούτε να δούμε πώ θα μπορέσουμε να, να, να δώσουμε συνέχεια στι ε, δεσμεύσει φανερών. Πάει όσον αφορά την, την, ανακεφα, την ανακεφαλαιοποίηση των ε, τραπέζων κλπ. Και, να μπορέσουμε τελικά να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τις ασύμμετρες κρίσεις, τα ασύμμετρα σοκ, τους ασύμμετρους κλειδονισμούς. Πολιτικές και άλλες στη συνέχεια της εξαπλής δέσμης. Δεν είμαι σίγουρος ότι πέρασε ξεκάθαρα το μήνυμά σας από την ε, μετάφραση. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι θέλετε σε σχέση με ε, αυτή την εξαπλήσμη. Γιατί, ας πούμε, τι, είπατε ε, για τον φόρο των χρηματοπιστωτικών πράξεων, συναλλαγών, όλοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν πάντως και να υπάρξει συνεργασία όλων για να προχωρήσουμε σε αυτά τα οποία τάξαμε ως προτεραιότητα που αναφέρατε. Α, εδώ μου λέει ο συνεργάτης μου. Μου λέει ο συνεργάτης μου που κατάλαβε την ερώτηση, δεν καταλαβαίνω αυτό που κατάλαβε ο συνεργάτης μου και εγώ. Η Κομισιόν θα πρέπει έχει τον γνωστικό ρόλο όσον αφορά τους στόχους για το έλλειμμα των κρατών Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επεξεργαστεί τις υποσχέσεις, τις δεσμεύσεις Ρομπάι. Ξέρω ότι δεν σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Συμπαθάτε με. Ε, καλά, στο τέλος του εξαμήνου θα, θα μας πείτε μεστότερα πράγματα. Τέλος πάντων. Ο Σον Κέλλη επανήλθε. Επομένως, ακόμη μια Ιρλανδική φωνή θα ακούσει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί είμαι μέλο τη Επιτροπή σας. Τακτικό, Τέλος πάντων. Καλώ όρισε ο Υπουργό. Θα σας πω ότι όταν αναλάβατε το Υπουργείο σας πριν από δύο χρόνια η Ιρλανδία βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού του πλευράς οικονομικής. Τώρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ανάκαμψης. Επομένως τώρα έχετε ευκαιρία να προωθήσετε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε που αναφέρατε για το εξάμεινο αυτό. Σε σχέση τώρα με την ύφεση και την κρίση πολλές φορές δικαίως κατηγορούμε τις, ε, του, τους φορείς πιστοληπτικής αξιοπιστίας και αξιολόγηση. Γιατί ξέρουμε τι κάνουν. Τι λέτε. Μήπως μπορείτε να διερευνήσετε, να προωθήσετε, τον έχουμε ένα τέτοιο οργανισμό αξιοπιστίας ευρωπαϊκό. Σκεφτείτε αυτό το επόμενο ξανά τόσο ώστε να έχουμε έναν ανταγωνισμό στην αγορά, ναι. να μην έχουν εκείνη η οίκη αξιολόγηση το μονοπόλιο. Να μην υποστούμε αυτές τις, τόσο φτωχές τους επιδόσεις όπως το παρελθόν. Και να κάνουν αυτά που κάνουν τα κυρία κράτη ένα τέτοιο οίκο αξιολόγηση όντω έχει υπάρξει, έχει πέσει ιδέα για να το φτιάξουμε, να έχουμε μια νέα τέτοια υπηρεσία. Και μόλις την περσμένη εβδομάδα τελικά υπήρξε συμφωνία. Να, έγινε πρόοδος επομένω. Εντάξει, φυσικά βέβαια είναι θέμα αξιοπιστίας πώς θα σταθεί, πώς θα λειτουργήσει αυτή η καινούργια υπηρεσία. Μπορεί να υπάρξουν κατηγορίες, επικρίσεις, ότι δεν θα είναι αμερόληπτοι. Κάποιες ε, θεωρούνται πιο άγγελες, κάποιες λιγότερο από αυτές τις του τους οίκους αξιολόγηση. Δεν έχει υπάρξει κανένα είδου ε, λύση προ το παρόν. Πρέπει να τι ενθαρρύνει να είναι πιο αμερόληπτε, πιο σωστέ να έχουν καλέ επιδόσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρος. Αυτό ισχύει και με τις εταιρείε που ασχολούνται με τα λογιστικά, με τους λογαριασμούς. Τέλος πάντων. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε και πιστεύω ότι όποτε χρειάζεται, όποτε θέλουμε να έχουμε κάποιο είδου τριμερή συνάντηση, να έρχεστε εσεί να μην έρχεται κανεί διπλωμάτη. Νομίζω ότι κάνουμε βήματα προόδου. Καλά τα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν προστριβέ μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά νομίζω ότι αυτή η Προεδρία νομίζω θα μα κάνει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, το ποτήρι μισογεμάτο. Και έτσι ελπίζω λοιπόν στο τέλο θα μα παρουσιάζετε επιτυχίες και που έχετε τόσα δύσκολα θέματα. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Και θα τα ξαναπούμε. Και με τους υπολείπους θα τα ξαναπούμε. Πότε, πω, πω. Α, όχι, όχι, δεν θα σας δω. Όχι, θα σας δω. Τέσσερις Δευτέρου στο Στρασβούργο. Το απόγευμα. Μακρά συνάντηση τότε για να ψηφίσουμε διάφορα. Θα ξαναπούμε μόνο στις 4 Φεβρουαρίου.